Ας αρχίσουμε, διότι πέρασαν 15 λεπτά, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. ορίζω τους πάντες. Όπως γνωρίζετε, μεταδίδεται και στο διαδίκτυο, όπως ε, χτες. Πριν πάμε στο εργαστήριο και τη συζήτηση περί διαφανείας, να σας πω κάποια πράγματα. Ελήφθησαν αποφάσεις εχθές από τους ε, συντονιστές και έχω καθήκον να σε ενημερώσω σχετικά. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις και την κατανομή τους, αποφασίσαμε ότι ΑΦΚΟ θα πρέπει να συντάξει γνωμοδότηση σχετικά με τα θέματα που εξεργάζεται η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για τη δημιουργία μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσης για δημοκρατία, κάτω δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Uh, Ζήτησε από Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να συμφωνήσει να γίνει γνωμοδότηση ε, για την έκθεση βάσει του άρθρου 54. Έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε αποκλειστικές αρμοδιότητες στον τομέα που έχουμε και να συμβάλλουμε στη σύνταξη της ε, εκθέσεως που ετοιμάζει η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και η γνωμοδότηση θα ανατεθεί στο ΕΛΚ. Επίσης ε, συζητήσαμε κατά πόσο αύκο θα πρέπει να μας γνωμοτήσεις για την απαλλαγή για τον προπολογισμό του 2014 και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Η συζήτηση όμως εστιάστηκε επί προετοιμασία γνωμοτήσεως για ε, την ενδεχόμενη θεσμική διάσταση της γνωμοδοτήσεως και ποιο είναι το πλαίσιο της απαλλαγής του προπολογισμού του Συμβουλίου αλλά θα ληφθεί απόφαση στην επόμενη συνεδρία. Συζητήσαμε επίσης τις νέες εκθέσεις που θα συνταχθούν από την ΑΦΚΟ τους επόμενους μήνες. Θα υπάρξει έκθεση για την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι δυνατότητες υπάρχουν, ποιες προκλήσεις. Εδώ οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες αλλά και το EFTD εξέφρασαν ενδιαφέρον. Θα ληφθούν αποφάσεις επ' την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Συμφωνήσαμε επίσης να ζητήσουμε έγκριση για σχέδιο εκθέσεως πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ε, πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, ποιες είναι οι θεσμικές συνέπειες στο νομικό πλαίσιο και αν καλυπτώμεθα από συνθήκες Αβώνας και πώς θα έχουμε μόνιμη δομή συνεργασίας. Δεν έχουμε τελική εκδοχή του τίτλου. Πιθανότατα η ΑΦΕΤ θα ζητήσει κάποια μορφή συνεργασίας από αυτού. Ο ε, θα είναι από την ομάδα του ΕΛΚ. Ζητήσαμε επίσης έγκριση για έκθεση για τις εφαρμοστικές διαστάσεις που είναι εκτός της, ε, των ποσοστώσεων των εκθέσεων θα αφορά την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης εντός του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα ανατεθεί στην ΓΚΟΕ η έκθεση. Επίσης συμφωνήσαμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει δυνατότητα και περιθώριο θα ζητήσουμε έγκριση για σχέδιο εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας για διάφορα συνταγματικά μοντέλα για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θα ξεκινήσει και μελέτη για το ρόλο του δημοψηφίσματος στα πλαίσια της διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πιθανότατα θα οργανώσουμε και ένα εργαστήριο από αυτού και ίσως τότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας. Θα ξεκινήσουμε με μελέτη και εργαστήριο. Αποστολές και ακροάσεις για το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνήσαμε να γίνουν δύο αποστολές. Αθήνα, που ανεβλήθη από το 2015 και Ισπανία και αυτό όμως πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα ανώτερα επίπεδα της, Ευρωπαϊκής, της Ιεραρχίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιθανότατα για το δεύτερο εξάμεινο θα εξτάσουν τη δυνατότητα να έχουμε Ουγγαρία, Σλοβακία και Πολωνία στο πρόγραμμά μας για αποστολές το δεύτερο εξάμεινο. Συζητήσαμε ακροάσεις συμφωνήσαμε να διεξαχθεί ακρόαση για την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ακρόαση για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κάτι που ήδη συζητήθηκε, να δούμε πού βρισκόμαστε, ποιε είναι οι συνέπειες μη ολοκληρώσεω της διαδικασία μέχρι τώρα και πώ να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη προκλήση στο μέλλον. Συμφωνήσαμε, διεξαχθεί ακρόση για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης στον ΟΗΕ, και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Επίσης συζητήσαμε το θέμα της Επιτροπής Αναφορών που μας έστειλε πληροφορίες που είπε ότι η Ιταλός πολίτης θα ήθελε το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι άνθρωποι σαν κι αυτόν που είναι ε, μέρος των ενόπλων δυνάμεων σε αποστολή ότι μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί στις ευρωπαϊκές εκλογές πρότεινα να το συζητήσουμε το θέμα μέσω των εργασιών που διεξάγονται για, την τροπο, για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Νόμου και να σας ενημερώσω ότι χθε επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι η μεικτή ακρόαση για την κοινή πολιτική ασφαλείας άφετ και αυκό μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας θα λάβει χώρα στις 13 Οκτωβρίου μετά τη συνθήκη Λισαβόνα. δηλαδή τι εννοούμε. Συνθήκη Λισαβόνα και πέρα, αυτό εννοούμε. Και από την ΑΦΚΟ θα έρθουν δύο πυρογνώμων. Ο καθηγητής Κουδράκος από το City University του Λονδίνου και ο κ. Στέφανος Σιλβέστρη, πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου ε, του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων της Ιταλίας. Αυτά συζήτησαν οι συντονιστές. Αν δεν έχετε σχόλια, αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή μας εγκρίνει αυτά που σας ανέφερα, δηλαδή τις αποφάσεις των συντονιστών. Θα θυμόσαστε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Φραντς Τίμερμαντς, έπρεπε να μεταβεί σήμερα στην Ιταλία. Αυτό στα πλαίσια του μεταναστευτικού προβλήματος, της κρίσης. Και δεν παρίσταται σήμερα, όμως θα διεξαχθεί συζήτηση παρόλα αυτά για τα θέματα που θέλαμε να συζητήσουμε μαζί του συζητήσεως με τους εμπειρογνώμονες που καλέσαμε και όλα αυτά στα πλαίσια της εκθέσεως Γκίγκολτ όπως αποκαλείται. Ο Σβέν Γκίγκολτ είναι συγγητής για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, για τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την ακαιρεότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο Σβέν θα αναφερθεί στο θέμα. Φιλοδοξία του είναι να έχουμε πιο συνεκτική προσέγγιση όσον αυτά τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα θεσμικά όργανα αυτής. Στηρίζουμε τη δουλειά του και θέλουμε να γίνει και πιο ορατή δουλειά του και γι' αυτό συμφωνήσαμε να δεξαχθούν μελέτες. Αυτές διεξήχθησαν τη Γενική Διεύθυνση IPOL, τη Διεύθυνση ε, Πολιτικής για Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικά Θέματα. Πρώτη μελέτη αφορά θεσμικές πτυχές της εκπροσώπησης διαφόρων συμφερόντων και μετά έχουμε τις δηλώσεις των οικονομικών συμφερόντων και ποιος έλεγχος επ' αυτών προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία. Είναι διαθέσιμες και έχουν διανεμηθεί αυτές οι μελέτες. Ο κ. Ντέβιτ Κοέν και ο κ. Ντόλμαιερ είναι οι συγγραφείς αυτών των εκθέσεων. Τους καλέσαμε να έρθουν και να κάνουμε εισαγωγή στη συζήτηση και να παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους και ο κύριος Γιάννος Μπέρτοκ είναι εδώ, επιφανής επαΐων επ' αυτών, επικεφαλής της, ακερι... της Διεύθυνσης για την Ακαιριότητα Δημοσίου Τομέα του ΟΣΑ. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες και έχουμε και τον Σβέν Γκίγκολτ. Να σε αποκαλέσω εμπειρογνώμονα, αλλά είσαι πολιτικός πιθανότατα, πολιτικός εμπειρογνώμων τέλος πάντων. Ας ξεκινήσουμε όχι με τον Σβέν αλλά με τον κύριο Γιάννος Μπέρτοκ, που είναι ο πρώτος που θα μιλήσει, από τον ΩΣΑ. Βλέπετε πολλά συμβαίνουν εκεί, περί, για τα θέματα της διαφάνειας, της ε, ακαιρεότητας κλπ. Και θα θέλαμε να μας κάνει μια παρουσίαση όσον αφορά το έργο που επιτελείται στον ΩΣΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να σας δώσω και την ε, σκοπιά των εθνικών κυβερνήσεων. Όσα, κατά την συντριπτική της πλειοψηφία, απαρτίζεται από κράτη-μέλη της Ένωσης, Έχουμε όμως και μέλη από την ΑΦΤΑ, τη βορειομεκανική δηλαδή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, από τον, από τον Ειρηνικό, Ιαπωνία, Κορέα και Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω αυτή την προοπτική και πρώτα να σας ε, αναφέρω τις ε, βασικές μας ε, ανησυχίες και τα βασικά μας μελήματα σε επίπεδο χωρών όσα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια βλέπουμε να υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Σήμερα δηλαδή, α, ωραία, ευχαριστώ, βλέπουμε και τις διαφάνειες τώρα, Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα φαίνεται να υπάρχει απώλεια εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το πλαίσιο και αν συγκρίνουμε ε, την κατάσταση πρώτης χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης υπήρχε κάποια αύξηση, αλλά βλέπουμε ε, μάλλον ήδη κάποια μικρή μείωση, αλλά τώρα βλέπουμε μεγάλη μείωση. 5% στα δίτρια των χωρών τόσα Κατά μέσο είναι η μείωση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς. Αν δούμε τις συσχετήσεις και το πόσα λεφτά ε, διασυνδέονται με ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, την ε, διαφάνεια θα δει κανείς ότι διαφάνεια καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πλέον στατιστικός σημαντική συσχέτιση. Από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι τα στοιχεία αυτά και στοιχεία του Γκάλοπ που δείχνουν την εμπιστοσύνη και ότι σχετίζεται με την ε, ανοιχτή διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένα σημαντικό μέρος της μελέτης στο ΩΣΑ είναι η άσκηση πιέσεων, το λεγόμενο lobbying. Και οι λομπίστες ε, και οι νομοθέτες θεωρούν ότι η διαφάνεια μπορεί να οδηγήσει και σε μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε εθνικό επίπεδο η διαφάνεια είναι μείζον ανησυχία και μέλημα, διότι βλέπουμε να συνάπτονται συμφωνίες και κλεισμένων των θυρών και ο στόχος είναι η αύξηση της διαφάνειας. Αν ε, επανέρχομαι, ξαναδούμε τις ε, τάσεις σε εθνικό επίπεδο, ε, σε εθνικών κυβερνήσεων, θα έλεγα ότι τα κράτη έχουν καταβάλει φανταστικές προσπάθειες. Έτσι θα αποκαλούσα. Οκτώ χώρες έχουν ε, εγκρίνει ε, νόμους ε, σε σχέση με τη διαφάνεια και το lobbying τα τελευταία 5-10 χρόνια. Για να κάνουμε μια σύγκριση με, τον προηγούμενο, με την προηγούμενη πεντηκονταετία, ήταν ο ίδιος ο αριθμός αυτός. Άρα, ό,τι έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια είχε γίνει τα τελευταία 50 πριν. Ε, θεαματικές προσπάθειες ε, και στην Ιρλανδία και πέρυσι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε αυτούς τους νόμους. Τώρα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και στη συστάση των συστάσεων του ΩΣΑ, η υλοποίηση σίγουρα είναι το αποφασιστικό στοιχείο. Και η υλοποίηση Ξεκινάμε την ευαισθητοποίηση, το awareness. Βλέπουμε εδώ την αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων και από τους νομοθέτες αλλά και από τους λομπίστες και μπορείτε να δείτε ότι δεν είναι τόσο γενικά αλλά ίσως εξατομικευμένα αυτά τα μέτρα που είναι πιο αποτελεσματικά. Η ενημέρωση, το briefing, η, τα εργαστήρια, η διαδικτύωση. αλλά άλλα κριτήρια όπως η πρόσβαση στις πληροφορίες, οι προσωπικές συμβουλές. Ανάλογα με το αν πρόκειται για τον νομοθέτη ή για τους λομπίστες, βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά τα, τα ποσοστά της αξιολόγησης των διαφόρων μέτρων. Ποια είναι λοιπόν τα διάφορα μέτρα. Έχουμε καταρχάς τον κώδικα συμπεριφοράς, Code of Conduct, οι λομπίστες πώς ε, εκτιμούν αυτόν τον κώδικα. Μιλάμε για μια αντιπροσωπευτική μελέτη που έγινε σε 100 ενώσεις ε, ομάδων άσκησης ε, πίεσης. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι κώδικες αυτής της συμπεριφοράς της δεν θεωρούνται αποτελεσματικοί. Δεν θεωρείται ότι παρέχουν κίνητρα, ούτε και αναγνώριση. Τώρα, περνάμε στη σκοπιά της συμμόρφωσης. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν θεωρεί ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές. Όπως και το άλλο σκέλος, η ανταμοιβή δεν λειτουργεί. Τι ενδιαφέρει και ανήσυχη πραγματικά Δύο πράγματα προέκυψαν από αυτήν την ε, μελέτη. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε revolving doors, τις περιστρεφόμενες πόρτες, δηλαδή μεταπίδεις από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ υπάρχουν ειδικά μέτρα, τα οποία εστιάζουν κυρίως στο πάνω-πάνω επίπεδο, στο εκτελεστικό δηλαδή, αλλά μέχρι στιγμής οι μισές μόνο χώρες του ΩΣΑ έχουν τέτοια μέτρα για τα ανώτατα εκτελεστικά στελέχη. Και αν δούμε τι μέτρα είναι αυτά, και δούμε την πλευρά των νομοθετών, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά γιατί είναι πάρα πολύ συχνό εδώ το φαινόμενο. για τα μέτρα που αφορούν αυτή τη μεταπίδηση από το δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Να σας δώσω ε, κάποια στοιχεία. Πριν από 40 χρόνια στο Κογκρέσο τον είπα μόνο το 4% των απερχόμενων ε, μελών του Κογκρέσου ε, πήγαιναν στον τομέα των λομπιστών. Όμως, στις τελευταίες εκλογές τρία χρόνια πριν είδαμε ότι οι μισοί, τις, οι μισοί γερουσιαστές έγιναν λομπίστες. Γιατί αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί τους προσλάμβαναν κυρίως και ο μισθός τους εξαρτώταν ακριβώς από την πρόσβαση που μπορούσαν να παρέχουν. Όταν άλλαζε ο εργοδότης, για παράδειγμα, υπήρχε μία μείωση του μισθού κατά πέντε ε, φορές. Έρχομαι στους λομπίστες τώρα και πάλι πολύ λίγες χώρες όπως βλέπετε έχουν μέτρα όταν ε, οι τέος λομπίστες ε, καταλαμβάνουν κάποιο κυβερνητικό αξίωμα. Βλέπετε και εδώ ε, το διάγραμμα που δείχνει ότι οι περισσότερες χώρες του ΩΣΑ δεν έχουν σχετικά μέτρα. Αν λοιπόν δούμε την πρακτική που επικρατεί, η μελέτη μας, η έρευνά μας έδειξε ότι φυσικά δεν υπάρχουν περιορισμοί. Όμως, αν δούμε πόσοι λομπίστες. διετέλεσαν κατά το παρελθόν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο αριθμός είναι υψηλός και αυξάνεται αυτή η πρακτική. Η δεύτερη ανησυχία είναι το λεγόμενο lobbying inside, θα το χαρακτήριζα, δηλαδή κάτι αδιαφανές εντελώς Δηλαδή οι λομπίστες και ιδίως τα, ανώτεροι, ε, τα ανώτερα στρώματα πλέον συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, ως συμβουλευτικές ομάδες. Πολύ λίγες χώρες είναι αυτές που έχουν περιορισμούς. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, όπως βλέπετε, τα τρία τέταρτα δηλαδή των χωρών του ΩΣΑ δεν έχουν περιορισμούς. Επομένως, ε, διευθύνονται σύμβουλοι, οι λομπίστε μέσα στα τρία τέταρτα, στα τρία τέταρτα των χώρων μπορούν να γίνουν εμπειρογνώμονε σε μια συμβουλευτική ομάδα. Τι μας λέει η τρέχουσα εμπειρία. Το 18% των λομπιστών είναι μέλη συμβουλευτικών ομάδων. Το βλέπουμε να γίνεται. Γιατί όμως αυτό αποτελεί πρόβλημα. Γιατί στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν μέτρα για την ε, ενημέρωση, για την πληροφόρηση ή για την δημοσιοποίηση πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη σύνθεση, τα καθήκοντα λοιπά αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, εν κατακλείδη, να τονίσω εκ νέου ότι η συμμόρφωση, δηλαδή η εφαρμογή, τα κίνητρα είναι σημαντικό στοιχείο. Δεν αρκεί η έγκριση κάποιων νόμων. Το θέμα είναι να δίνονται κίνητρα, να παρέχονται εργαλεία για την εξασφάλιση ε, της ε, συμμόρφωσης. Δεύτερο, σχετική έλλειψη δεδομένων για τον αντίκτυπο για το τι αποδίδει και πώς. Δηλαδή, ποια εργαλεία μπορούμε να θεωρήσουμε αποτελεσματικά, ποια εργαλεία λειτουργούν, ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος. Τρίτον, συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφάνεια, για την ακαιρεότητα. Αν δεν υπάρχει αλληλοϊποστήριξη μεταξύ των διαφόρων μέτρων ε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και εδώ σας δίνω κάποιες ε, πληροφορίες για τις απόψεις των ε, μελών ομάδων πίσης, ομάδων πίσης και των νομοθετών για το τι είδους πληροφορίες θεωρούν σημαντικό να δημοσιοποιούνται πολύ σημαντικό είναι η χρηματοδότηση εκλογών και χρηματοδότηση κομμάτων, για παράδειγμα. Περισσότεροι νομοθέτες, το 84% θεωρούν ότι είναι μείζον το ζήτημα αυτό. Λόμπινγκ και σχέση με χρηματοδότηση κομμάτων. Ένα άλλο θέμα είναι ποιος καλύπτεται, ποιος διέπεται από τους κανόνες για το λόμπινγκ. Υπάρχει αίσθηση ότι υπάρχει ένα πιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και βλέπετε κάποια μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί, κάποια κατόφλια για παράδειγμα ή κάποια έγγραφα ε, που δημοσιοποιούνται κτλ. Και τέλος, κίνητρα. Στον νόμο Βασίλειο για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται όλο και πιο συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα της οικονομικής συμπεριφοράς. Έχουμε το θέμα της, διαφα... της ε, γραφειοκρατίας. Ένα μέτρο λοιπόν είναι η καταχώρηση και υποβολή αναφορών. «30 λεπτά διαρκεί περίπου η καταχώρηση Καταλαβαίνω την πλευρά βέβαια των ανθρώπων αυτών, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σίγουρα μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας. Έχω φέρει όμως και δύο-τρία γλυκά αντίγραφα και κάποια βασικά ε, σημεία αυτής της έρευνας. Σας ευχαριστώ. Ε, thank you, Mr. Um... Ε, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. αντικαθιστώ την Τανούτα, μάλλον επειδή είμαι ο πρεσβύτερος, άλλο λόγο δεν βλέπω. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο David Κιούν, ο οποίος έχει συντάξει μια μελέτη για σταγματικές και αντισταγματικές πτυχές και την εκπροσώπηση από το τμήμα του Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από το London Business School, το Max Planck, έχει διδακτορική διατριβή για business lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τιμηθεί από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας το 2015. Είχε την έδρα Κορδέλα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας 2008-2009. Είχε ε, ήταν επισκέπτης ε, στο Kennedy School του Harvard. Έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με ρυθμιστικά δίκτυα και ευρωπαϊκό λόμπι. Έχετε το λόγο 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Μακροσκελής η παρουσία σας. Όντως 20 χρόνια έχω αφιερώσει τα λόμπι. Νομίζω ότι αυτό αρκεί ως εισαγωγή. Ολοκλήρωσα μια μελέτη των λεγόμενων revolving doors στις Βρυξέλλες, των ε, κυκλικών θυρών, αν και τις ονομάζουμε μάλλον κυλιόμενες ε, θύρες και όχι κυκλικές. Αλλά μάλλον αυτό αντιστοιχεί περισσότερο στην πραγματικότητα. Ε, η σημερινή παρουσίαση λοιπόν προκύπτει μετά την έκθεση που θα έχετε δει φαντάζομαι δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα έγινε για λογαριασμό της Επιτροπής των Σταγματικών Υποθέσεων και στόχο έχει τη μελέτη των το, του ρόλου των λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το, τη λειτουργία του, λόμπι, του Μητρώου Διαφάνειας, ε, τα δεδομένα διαπίστευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανάλυση ακροάσεων και μια μελέτη μοναδική, νομίζω μοναδική, επί των Ευρωβουλευτών. Ήρθαμε σε επαφή με πολλούς από εσά, με ερωτηματολόγια από τον ε, Σεπτέμβριο τον, στον Απρίλιο του 2015 με μια καλή ανταπόκριση και αποτέλεσμα μια μελέτη 400 σελίδων για την οποία μπορώ να σας δώσω κάποιες ε, περιορισμένες μόνο, μια επισκόπηση μόνο, αλλά όποιος θέλει πολύ ευχαριστώ να συνομιλήσουμε λεπτομερέστερα μετά. Καταγράφουμε λοιπόν τον αριθμό των ομάδων ε, συμφερόντων, την κατανομή τους, την ε, ποικιλία τους, την ένταση τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάζουν με την παρουσία τους. Ποιος δηλαδή, που ασκεί εκπροσώπηση από ομάδες πιέσεις, πιέσεως και τι είδου συνέπειες μπορεί να προκύψουν από αυτές τις, ε, τη διαφορετική ένταση της πίεσης των ομάδων πιέσεων. Ε, το βαθμό στον οποίο μπορεί να τροποποιηθεί, η επιλογή μιας πολιτικής, η διαφάνεια, η λογοδοσία και Θέλησαμε να δούμε επίσης ποιος μιλούσε σε ευρωβουλευτές, σε τι ε, συχνότητα και επίπεδο και γιατί δέχονταν οι ευρωβουλευτές να συνομιλήσουν με τις ομάδες πιέσεως και τι συνέπειες μπορεί αυτό. 20-30 ερωτήσεις λοιπόν ε, που αναλύουν πολλά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από τις διάφορε επιτροπές. Πρώτα λοιπόν, Έχουμε κυρίως την παρουσίαση στον πρώτο πίνακα της πιστοποίησης ανάλογα με τις επιτροπές για την περίοδο 2012-2014. Το πρώτο, η πρώτη διαπίστωση να κοιτάμε τα στοιχεία αυτά βλέποντας τις ε, οργανώσεις που βρίσκονται μέσα στο Κοινοβούλιο, βλέπουμε ότι κατά 50% είναι εσωτερικές, αυτό που ονομάζουμε in-house. 27% μη κυβερνητικέ οργανώσεις και 18 ε, επιχειρήσεις. Με το Μητρό Διαφάνειας η σύγκριση δείχνει ακριβώς τα ίδια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 49% in-house, 26% μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εκεί Πράγμα το οποίο είναι ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη μπορεί να εξηγείται από το γεγονό ότι χρηματοδοτεί με κυβερνητικέ οργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδα δε επιχειρήσει ήταν κάπου στο 12% λίγο χαμηλότερο από το Κοινοβούλιο. Βλέπουμε λοιπόν μια ομοιότητα ω προ την γενική εκδήλωση του ενδιαφέροντο, αν όχι στα, συνολ... στα επιμέρου ποσοστά, πάντω στα σύνολα εκπροσώπηση Κοινοβούλιο Επιτροπή. Θέλησαμε όμω να δούμε και την κατανομή ανάλογα με τους τομείς της πολιτικής. Και έτσι κάνουμε την, ε, σπάμε τα στοιχεία ανάλογα με τις, ευρωπαϊκές, με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε αν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά σε σχέση με το είδος της πολιτικής. Κοινοβούλιο και Επιτροπή πάντα. Από τα γραφήματα αυτά που βλέπετε, οι οικονομικές όπως τα λέγαμε ομάδες εργασίας, η πιέσεως καλύτερα, ε, εστιάζονται στις πολιτικές στις επιτροπές που ασχολούνται με την εσωτερική αγορά, γενικά οικονομικού ενδιαφέροντος με θέματα ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, ε, περιβάλλον, καταναλωτές. Εδώ έχουμε σαφέστατη παρουσία, εκπροσώπηση και επιρροή των οικονομικών ομάδων από τις ε, in-house της εσωτερικής δραστηριοποίησης όπως λέγονται. και αυτό βέβαια εξήγεται και το γεγονός ότι επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, δηλαδή την ε, δυνατότητα μια πολιτική που επιλέγεται από το Κοινοβούλιο να φέρει αποτελέσματα. Αυτό επίσης εξηγείται και από την διαδικασία των πρώτων αναγνώσεων και την συνεργασία για να περάσουν τα θέματα σε πρώτη ανάγνωση. Ω κοινοβούλιο δηλαδή, αν θέλει κανείς να συνεργαστεί με την Επιτροπή, πρέπει να έχει και την τεχνική υποστήριξη, την τεχνογνωσία, για να μπορέσει να έχει επιχειρήματα σε ένα πιο ισότιμο ε, πεδίο γνώση του τομέα της πολιτικής. Είναι μη κυβερνητικέ οργανώσει, αντίστροφα, είναι πιο ορατέ τη περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα επιτροπές εκείνες που έχουν πιο πολύ αναδιανεμητικές δράσεις πολιτικών ελευθεριών, ανάπτυξης, πολιτισμού και πάλι ε, με την νομοποίηση και νομοποίηση της ενημέρωσης με βάση την οποία θα λάβει κανείς πολιτικές αποφάσεις δηλαδή προσπάθεια από το Κοινοβούλιο να έχει στο δυνατόν περισσότερη γνώση, επικοινωνία, επαφές με ομάδες συμφερόντων και ε, εκπροσώπους, αντίστοιχα ε, σε ισότιμο επίπεδο με αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να έχει τις γνώσεις για να λάβει αποφάσεις. Άρα βλέπουμε ότι είναι πιο ε, διατεθειμένες να ακούσουν ευρύτερη κλίμακα εκπροσώπων συμφερόντων οι επιτροπές αυτές, ανάλογα βέβαια και με την ε, κατανομή βλέπουμε τι είδους κατευθύνσεις έχουν τα συμφέροντα που εκπροσωπούνται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Άλλες πολιτικές διαδικασίες επίσης βλέπουμε να ε, φέρνουν αλλαγές. Φέρει η διαδικασία της ίδιας πρωτοβουλίας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον από τα λόμπι και η υποδοχή από το Κοινοβούλιο. Θετική λοιπόν αντιστοίχηση βλέπουμε σε σχέση με τις ε, ομάδες ε, συμφέροντος κατά την εισαγωγή ή από την εισαγωγή της διαδικασίας ε, ιδίας πρωτοβουλίας, αλλά αντίστοιχα και σε άλλες διαδικασίες και ιδιαίτερα όπως είπα και στην πρώτη ανάγνωση, και επίσης βλέπουμε ότι ε, καθώς είναι όλο και περισσότερες οι πρώτες αναγνώσεις, θέλοντας οι βουλευτές να ξέρουν ότι μπορούν να παρακολουθήσουν ε, με τις γνώσεις τους ε, τα θέματα και να τα υποστηρίξουν, ίσως έχουν μεγαλύτερη επικοινωνία με τις ομάδες συμφερόντων. Και υπάρχει και άλλη μία αντιστοίχηση, παρουσία αντίστροφη, το ότι δείχνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ενδιαφέρον στις διαδικασίες που μπορούν να κλείσουν σε πρώτη ανάγνωση. Είπα και οι ίδιες πρωτοβουλίες που έχουν πολιτικό χαρακτήρα και θέλει το Κοινοβούλιο να ορίσει το πολιτικό θεματολόγιο και να το επηρεάσει περισσότερο, νομιμοποιεί κατά κάποιον, και νομιμοποιήσει κατά κάποιον τρόπο την παρουσία του στην ε, πολιτική σκηνή της Ευρώπης και σε σχέση με την κοινή γνώμη, πάλι εξηγεί και δικαιολογεί την παρουσία των ε, λόμπι. Κάτι που δεν έχω εκθέσει εδώ είναι οι φύλακες πολιτικής που έχουμε αναλύσει. Επιμέρους δηλαδή ιδιώτες επιχειρήσεις ε, και συγκεκριμένα σε ποια επιτροπή προσήλθε ο καθένας ή πόσες φορές προσήλθε ο καθένας ή η καθεμία ομάδα συμφερόντων. Δηλαδή πόσες φορές ακούστηκε η καθεμια ομαδα συμφεροντων δηλαδη ε, ποσες αυτών των ε, εκπροσώπων. Και εδώ βλέπουμε θύλακες γύρω από τις οικονομικές βιομηχανικές επιτροπές με τα ίδια άτομα και εκπροσώπηση, ή ομάδες συμφερόντων ε, γύρω από τις ίδιες επιτροπές. Ο θύλακας για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αφορούσε πάλι τα σταγματικά, την εξωτερική πολιτική κτλ. Με σημαντική παρουσία αυτών των παραγόντων στη συνεδριάση των επιτροπών. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να ε, σας καταπλήξει, αλλά πάντως δείχνει ότι οριμάζει στη διαδικασία αυτή το κοινοβούλιο, είναι ότι φαίνεται να έχει μια πιο γενική επισκόπηση τη αντιμετώπιση της πολιτικής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο τεχνική προσέγγιση, καθώς είναι συνομοθέτης όλο και περισσότερο, διατυπώνει δηλαδή, συμμετέχει στη διατύπωση της πολιτικής. Με συνέπεια αυτό επιτροπές του Κοινοβουλίου να προσεγγίζουν ως προς την πολιτική της Γενικής Διευθύνης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάναμε την αντιστοίχηση και ναι μεν υπάρχουν διαφορετικές, ε, διαφορετικές ως προς αριθμούς ομάδες συμφερόντων ε, εδώ και εκεί, αλλά ε, ως αναλογίες, οι αναλογίες παρουσίας αυτών των ομάδων στις Γενικές Διευθύνσεις αφενός και στις Επιτροπές του Κοινοβουλίου Αφετέρου ήταν ε, ο ίδιος όπως είπα και νωρίτερα, κάπως λιγότερες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έρχονται στο κοινοβούλιο, σχέση με αυτές που έρχονται στην Επιτροπή. Ίσως αυτό θα ήταν το αντίθετο από ό,τι περιμέναμε. Αφού θεωρείται ότι το κοινοβούλιο είναι η φωνή τη κοινωνία των πολιτών και είναι ανοιχτό στο ευρύτερο κοινό κτλ. Αλλά από την άλλη, αν δούμε τι είδου πόροι και τι δυνατότητα μπορεί να έχει ε, για κινητοποίηση η συγκέντρωση ενδιαφερομένων και ενδιαφέροντος, αυτό εξηγεί την υποεκπροσώπηση. Δηλαδή οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις προσπαθούν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους ε, και, τους, και την παρουσία τους ε, στον ε, πρωταγωνιστή της πολιτικής διαδικασίας, δηλαδή την Επιτροπή και ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε στη συνέχεια κάποιες συστάσεις για το τι άλλο θα μπορούσε να κάνει το Κοινοβούλιο για να ε, αλλάξει αυτές τις ισορροπίες. Πολλά άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε μέσα στην έκθεση. Δεν είχαμε βέβαια ε, νομοθετική απεικόνηση ίχνος της παρουσίας ακριβώς για λόγους χρονικούς, αλλά πάντως βλέπουμε με πολύ ενδιαφέρον τα θέματα που προκύπτουν από το Μητρό Διαφάνειας, από, από τα στοιχεία διαπίστευσης και από τα στοιχεία τα σχετικά με τις ακροάσεις. Κάτι άλλο τώρα. Πώς έχουν ε, επαφή, επικοινωνία με τους ευρωβουλευτές ε, τα συμφέροντα και αυτό το λέω με ιδιαίτερη έμφαση γιατί νομίζω δεν υπάρχει άλλη μελέτη και πάντως συστηματική μελέτη που να έχει παρακολουθήσει ολόκληρο ένα κοινοβούλιο ή ολόκληρη ή μια γερουσία ως προς την πρόσβαση των ομάδων πιέσεως ή λόμπι στα μέλη τους. Όλα αυτά τα δίνει η έκθεσή μας λοιπόν θα δώσω, θα δώσω κάποιες ε, γενικές εικόνες καταρχάς. Η μελέτη μας δείχνει και τα αναμενόμενο φαντάζομαι ότι οι ευρωβουλευτές είναι όλοι ε, δεκτικοί, ανοιχτοί στις ομάδες πιέσεως σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων πιέσεως, ε, δημόσιες σχέσεις, εταιρείε δικηγορικές, στο βαθμό βέβαια που αυτές ε, καταγράφονται, ακόμη και ομάδες θρησκευτικέ που ίσως θεωρούνται λιγότερο θεμητές και πιο αμφισβητήσιμες, τουλάχιστον από τις απαντήσεις που λάβαμε, εκπροσωπήσεις περιφερειών και το καθεξής. Ο ρόλος των κρατών μελών επίσης στο lobbying στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλη σημασία και καταγράφεται. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και οι εσωτερικέ ομάδε ομάδες in-house είναι οι πιο συνήθει και ευάριθμε και πολυάριθμες. Πιο δραστηριε φαίνονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ενώ είναι λιγότερε δηλαδή μπορεί να έχουν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση ω προς τους τομείς του οποίου έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προτίμηση. Και όπω είπα και νωρίτερα, μεγάλο είναι και η δραστηριοποίηση των κρατών μελών σε όλη τη διαδικασία πολιτικής, όχι μόνο στα πολιτικά δηλαδή στάδια χάραξης πολιτικής. Στον κύκλο χάραξης πολιτικής, ε, ιδιαίτερα στην στη διαδικασία των τροπολογιών και τη ψηφοφορία σε ολομέλειες ε, βλέπουμε εντατικοποίηση της δράσης, αλλά και σε άλλες ε, φάσεις πιο πρώιμες, με κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, εκπρόσωποι συμφερόντων και ακόμα και στη φάση ε, πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσίαση των προτάσεών της βλέπουμε να εντατικοποιείται η παρουσία του. Ιδιαίτερα δε στην πρώτη ανάγνωση εντατικοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία αυτή και οι ευρωβουλευτές βλέπουμε να συνεργάζονται πολύ, σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο με τις ομάδες συμφερόντων από ό,τι συνέβαινε σε προηγούμενες θητείες του Κοινοβουλίου. Αυτό για μένα ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές των διαπιστώσεων, δηλαδή σε πρώιμο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας και ακόμα και στη φάση της προετοιμασίας και κατάθεσης των προτάσεων της Επιτροπής βλέπουμε στενή συνεργασία των λόμπι με το Κοινοβούλιο. Η παρούσα γραφική παράσταση δείχνει επαφές στις οποίες έχουν ε, προχωρήσει οι ομάδες συμφερόντων ε, στα διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, πολιτική, χάραξης πολιτικής. Σε ποιο στάδιο, ανάλογα με τον τομέα της πολιτικής, ανάλογα με το είδος της ε, ομάδας συμφερόντων και φαίνεται ότι επανέρχονται και επαναλαμβάνουν διαρκώ το μήνυμά του για να αποτυπωθεί καλύτερα στον Ευρωβουλευτή. Βλέπουμε κάποιους θύλακε όπου οι ιδιαίτερε ομάδες συμφερόντων φαίνεται να έχουν πιο ισχυρή φωνή, η μεγαλύτερη απήχηση. Δημόσιες ε, σε θέματα ε, δημοσίου δικαίου, χάραξη πολιτικη τα νομικά ζητήματα. Είναι πολύ πιο εμφανής η παρουσία τους. Γιατί, γιατί εκπροσωπούν πολλά διαφορετικά συμφέροντα συχνά είναι πρωταγωνιστές και μπορούν, όπως άλλωστε και με τα think tanks, να βρουν τις προτάσεις σύμπτωσης, σύγκλησης που θα επιτρέψουν την πρόσκοπτη προόδο ενός νομοθετήματος στη διαδικασία την νομοθετική γιατί θα μπορέσουν να συμφωνήσουν οι συνομοθέτες. Νομίζω ότι αυτή η παρουσία τους τις καθιστά σε πιο πρώιμο στάδιο ορατές. Ενώ οι επιχειρήσεις με κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. φαίνεται να είναι πιο ορατές στη διαδικασία της διατύπωσης όπως την ονομάζουμε γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν στο τέλος τα νομοθετήματα ή στους οποίους απευθύνονται τα νομοθετήματα και γι' αυτό επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν νομοτεχνικά τα κείμενα. Και όπως είπα αυτό συμβάλλει και στην ε, αποτελεσματικότητα και την ομοποίηση του αποτελέσματος. Αυτό βέβαια γεννά το ερώτημα το πώς μπορεί ένας ευρωβουλευτής να ε, κρίνει όταν είναι μεγάλη η ε, διαφοροποίηση των θέσεων που εκφράζονται, δηλαδή δεδομένων των, δεδομένης πολυφωνίας μπορεί να εκφράζεται προς, μια, προς πολλές κατευθύνσεις από τα λόμπι της μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις. Πώς θα κρίνει δηλαδή ένας ευρωβουλευτής. Και κάτι άλλο, όπως είπαμε, κράτη-μέλη συμμετέχουν διαρκώς στη διαδικασία. Ε, η προτίμηση αυτό που ρωτήσαμε του ευρωβουλευτέ ήταν πώς βλέπουν την επιρροή των ε, ομάδων συμφερόντων. Η απάντηση που λάβαμε πρώτα απ' όλα ήταν ε, παρουσία των κρατών ως νομιμοποιημένων. Στη συνέχεια μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ομάδων που έχουν την νομοποίηση και σε τρίτο στάδιο ανάλογα με τη δράση. Κάποιες ομάδες θεωρήθηκαν ε, λιγότερο, αποτελεσματικές, λιγότερο νομοποιημένες και λιγότερο αποδεκτές ως συνομιλητές όπως ε, αυτές που έχουν να κάνουν με την ε, χάραξη, που ενδιαφέρονται μάλλον για τη χάραξη πολιτικής κτλ. Στα ερωτηματολόγια μας ρωτάμε τι σημαίνει περισσότερη πρόσβαση, τι απαιτείται για να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση, τι μπορείτε να προσφέρετε. Και βλέπουμε από μεγάλο φάσμα των ομάδων ε, συμφερόντων και την προσφορά τεχνογνωσίας αλλά και πολιτικής ενημέρωσης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πολιτική τοποθέτηση και πολιτική φωνή και επιτυχάνουν περισσότερο εκείνες οι οποίες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα τεχνογνωσίας και πολιτικών επιλογών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή με την αντίληψη του τι είναι καλό για την Ευρώπη στο συνολά της, αλλά και για το εθνικό επίπεδο, δηλαδή κράτη-μέλη πιο επιτυχείς ήταν αυτές οι οποίες μπορούσαν δηλαδή σε όλους τους διάβλους επικοινωνίας να προσφέρουν πληροφορίες, όχι μόνο μια τεχνική έκθεση δηλαδή, ένα τεχνικό δελτίο, αλλά και το ε, πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούσε να τοποθετηθεί στην ευρύτερη πολιτική στα ευρύτερα πολιτικά δεδομένα. Σε σχέση με την στάση του σέρατε της διαφάνειας Οι απαντήσει ήταν ότι θεωρούσαν αποδεκτό το να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, μαζί τους οι ομάδες συμφερόντων. Ε, το θέμα της διαφάνειας ωστόσο θελήσαμε να δούμε εμείς εάν το Μητρό Διαφάνειας βελτιώνει τη συμπεριφορά και την εκπροσώπηση. Εάν, λοιπόν, στο ερώτημα εάν βελτιώνει τη συμπεριφορά των ομάδων συμφερόντων, περίπου το 60% συμφωνεί. Ε, Κάποιοι, κάπου στο 30% διαφωνούν με αυτή την ε, διαπίστωση. Πιο ασαφές είναι όμως, ε, πιο σαφής είναι η απάντηση στο ερώτημα εάν περιορίζεται η ε, μη ορθή συμπεριφορά των ε, ομάδων συμφερόντων χάρη στο Μητρό Διαφάνειας. Και εκεί είναι μοιρασμένες απαντήσεις. θα δείτε σε επόμενε δύο ερωτήσει και αυτό είναι σχετικό και με την προηγούμενη παρουσίαση, θα το συζητήσουμε μετά. Η ερώτηση παριθμό 3 λοιπόν αναφέρεται στο αν βελτιώνεται η διαφάνεια. 78% λένε ότι είναι πιο ανοιχτή και διαφανή στη διαδικασία στις Βρυξέλλες και εγώ που έχω μελετήσει και αλλού την παρουσία των λόμπι μπορώ να σα πω ότι όντω ε, αξίζουν συγχαρητηρίων οι Βρυξέλλες για την παρουσία τη διαφάνεια σε σχέση με τα λόμπι. Αλλά εάν υπάρχει περίπτωση να ε, συμπεριφερθούν κατά τρόπο εσφαλμένο και αν αυτά η παράβαση των καρών θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τη Μητρό ε, Ήταν, η απάντηση σε αυτό ήταν ότι ήταν επερκής. Και επίσης το εάν είναι χρήσιμο το Μητρό, Μητρό, και για τις ίδιες ομάδες ε, συμφερόντων. Και εκεί πάλι οι θετικές απαντήσεις ήταν περισσότερες. Ήταν κοντά στο 66%. Κάναμε λοιπόν μια σειρά από αναλύσεις για το τι ε, ομάδες συμφερόντων είναι παρούσες, τι κάνουν, σε ποιο βαθμό. Αλλά στην συμπεριφορά τους, την ομότυπη ή παράτυπη, είχαμε λιγότερη δυνατότητα να αξιολογήσουμε. Στα συμπεράσματα λοιπόν και τις συστάσεις μας, πολύ περιορισμένες γιατί δεν μπορούσαμε να εκθέσουμε τα πάντα μέσα 15 λεπτά, Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη δραστηριότητα των δημοσίου συμφέροντος ομάδων που το περιβάλλουν, ιδιαίτερα σε επιτροπές που έχουν περιορισμένη δραστηριοποίηση, με τις διαβουλεύσεις, με περισσότερη παρουσία και ποικιλία της εκπροσώπησης των θεμάτων και ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία χάραξης πολιτικής. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί, το, να ενισχυθεί η υπηρεσία έρευνας και τεκμηρίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξέρουμε ότι ως μονάδα έχει επεκταθεί αλλά αυτό που θα ήθελα να σημειώσω εγώ είναι ότι θα ήταν καλό να υπάρχει περισσότερη υποστήριξη απευθείας από τη γραμματεία της στους συντάκτες, στους ε, ε, συντάκτες νομοδοτήσεων και στους συγητές ε, των εκθέσεων για να μπορούν καλύτερα οι ευρωβουλευτές να ε, επεξεργάζονται την, ε, το μεγάλο όγκο των πληροφοριών που φτάνουν στο γραφείο τους η δυνατότητα δηλαδή για περισσότερη ανάλυση των αρχικών δεδομένων αντί για δευτερογενές υλικό που περνάει μέσα από τη διαβούλευση. Και αυτό νομίζω δίνει καλύτερη αντίληψη για τον Ευρωβουλευτή και της διαδικασίας ιδίας πρωτοβουλίας και γενικά όλου του όγκου της ε, νομοθεσίας περνάει μέσα από την πρώτη ανάγνωση μόνο. Επίσης θα πρέπει τόσο ε, το προσωπικό όσο και γενικά όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ευαισθητοποιηθούν ως προς στην ε, πρωτοβάθμια επικοινωνία με ομάδες συμφερόντων, ε, σε περίπτωση δηλαδή παράβασης των κανόνων ε, να υπάρχουν αυστηρότερες κυρώσεις και το καθεξής, να πιεστούν οι ομάδες να τηρούν τους κώδικες συμπεριφοράς πιο σωστά. Επίσης, συγκεκριμένες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιων ομάδων. Εμείς μπορέσαμε πολύ λίγο να ανοιχνεύσουμε τον αντίκτυπο των, των ε, ομάδων πιέσεων αυτών. Ενώ είχαμε ακούσει πάρα πολλά, το ίχνος τους δεν το είδαμε στην πράξη και έχουμε πολύ λίγους ευρωβουλευτέ όπου έχουμε καταγράψει μάλιστα σε πίνακα με ανώνυμα στοιχεία. Πολύ λίγοι ήταν οι ευρωβουλευτές ε, που ε, ομολογούν το νομοθετικό ίχνος των ε, ομάδων συμφερόντων και νομίζω ότι αυτό θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπαμε σε ποιο βαθμό εισακούστηκαν τα σχόλια των ομάδων συμφερόντων. Επίσης θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνεια και νομοποιήσει το Κοινοβούλιο διαθέτοντας ε, στο κοινό τις πληροφορίες και τη διαπίστωση ή την καταχώρηση στο Μητρό πρόσβαση και τρόπος παρουσίασης δηλαδή των δεδομένων κυρίως μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο τα δεδομένα πιστοποίησης να ε, γίνουν ορατά σε πίνακες ε, ή μάλλον σε αρχή HTML όπως παρουσιάζονται δεν είναι καθόλου εύχριστα και δεν μπορεί το κοινό να έχει πρόσβαση ευχαίρει. Επιπλέον σε σχέση με τα ιδιαίτερα συμφέροντα, οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσα από τα στοιχεία της πιστοποίησης κτλ. Θα πρέπει να είναι πιο σαφή ώστε να βλέπουμε ποιος συμμετέχει, ποιες ομάδες ε, συμφερόντων πηγαίνουν σε ποια επιτροπή ή επικοινωνούν με ποια Γενική Διεύθυνση Επιτροπής. Θα ήταν καλό να δούμε πού υπάρχει διπλή προσέ, διτή προσέγγιση, γιατί μια, ομα, μια επιχείρηση δεν έρχεται πάντα ως επιχείρηση, έρχεται ως ένωση πολιτών ως ε, δικηγορική εταιρεία, συνεργαζόμενοι και με μη κυβερνητική οργάνωση επίσης. Εγώ νομίζω όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απέτηση να καταγράφονται όλα τα επιμέρους συμφέροντα και η παρουσία τους του κάθε ενός και σε άλλους χώρους, ώστε να μην υπάρχει αυτή η διπλή, τριπλή, καταγραφή της ίδιας φωνής. Και κάτι ακόμη, συμπερίληψη σε ένα βαθμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα συστήματα αυτά θα βοηθούσε περισσότερο να αντιληφθούμε την ε, πίεση και την παρουσία των λόμπι στη διαδικασία παραγωγής αποφάσεων και πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό και έχω πει και σε προηγούμενη περίσταση ότι θα ήταν καλό να μην απευθύνουμε, να μην διατυπώνουμε ευχές που μπορεί να έχουν αντίξω αποτελέσματα, γιατί είναι άλλο το να πούμε ε, ποιο πρόσωπο, ποιος ιδιώτης εμφανίστηκε και μίλησε και άλλο το να ξέρουμε ποιος επηρεάζει τα κράτη-μέλη ιδιαίτερα. Και όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα, υπάρχει τεράστια απόκληση, ποικιλία και διαφορά πολιτικής βούλησης στα κράτη-μέλη στο θέμα αυτό και γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολο να ζητήσουμε ε, την ανείχνευση της παρουσίας των λόμπι μέχρι τη, τα πρωτή προτεύσεις των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ, αλλά αν θέλετε πολύ ευχαριστώ να τα πούμε και στο καφέ μετά. Ευχαριστώ καθηγητά Κοέν. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ο κ. Μπρόμαια μπορεί να ακολουθήσει. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Καθυστερήσαμε λίγο. Αλλά δεν θέλω να σας στερήσω από το χρόνο ομιλία σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρουσιάσουμε λοιπόν αυτό το πόνημα που ετοιμάσαμε από Μάιο μέχρι Ιούνιο φέτος. Βασικά να δούμε το δεντρολογικό κώδικα των μελών του Ευρωκοινοβουλίου Εξετάσαμε λοιπόν πέντε βασικές συνιστώσεις του δεντρογικού αυτού κώδικα, τους κανόνες, προσανατολισμό, πώς συμμορφώνεται κανείς με τις απαιτήσει, έλεγχος όσον αφορά τις δηλώσεις συμφερόντων, κυγώσεις και πώς ε, αναφέρονται διάφορες επιχειρήσεις. Θα αναφερθώ στο ευρύτερο πλαίσιο και μετά θα παρουσιάσω τα συμπεράσματα και συστάσεις. Τι εξετάσαμε εξετάσαμε το λογικό κώδικα για τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, πολύ προσεκτικά. Μα ζητήθηκε αυτό διότι στι αρχές του έτου συμμετείχαμε σε μια μεικτή ακρόαση για τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την ακαιρεότητα όπου παρουσιάσαμε έρευνα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από εμά όσον αφορά τον Λογικό κώδικα των μελών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάναμε. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί όταν μας ζητήσατε να εξετάσουμε αυτό τον κώδικα, τον εντολογικό, τον κώδικα συμπεριφοράς. Είχαμε την ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχαμε την υπόθεση Γκρέκο ε, και εκεί διεξήχθη μια έρευνα όσον αφορά των συστημάτων ελέγχου ακεραιότητα σε όλα τα κάτι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπη. Είχαμε και συμμετοχή 20 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσης, πολύ υλικό που εξετάσαμε, υπήρξαν πολλές προσεγγίσεις για να εξετάσουμε τα θέματα αυτά εντός των διαφόρων νομοθεσιών των κρατών μελών, διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ προσεγγίσεων βασίζονται σε αξία, βασίζονται σε κανόνες, συνδυασμό των δύο, ούτω ώστε να υπάρχει η ακαιρεότητα αυτή που θέλουμε με βάση ηθικές αξίες και προδιαγραφές. Γρήγορα τώρα σας δίνω μια επισκόπηση. Οι πρώτες διαφάνειες δείχνουν ένα χάρτη σε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπουμε τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του Κοινοβουλίου. Βλέπουμε τις χώρες, τις σκοτεινές, με σκοτεινό γαλάζιο όπου το Γκρέκο δεν έκανε συστάσεις. Χώρες όπου η ομάδα Γκρέκο εν γέννη βρήκε ότι αυτά που ίσχυαν όσον αφορά τους κανόνες μπορούν να θεωρηθούν να αποτελούν καλή πρακτική και ότι λειτουργούν και με ανοιχτό γαλάζιο είναι οι χώρε όπου το Γκρέκο έκανε συστάσεις και χρειάζονται βελτιώσεις. Και το Γκρέκο αναφέρει τι πρέπει να γίνει. Μια χώρα είναι γκρίζα, η Δανία, διότι έχει εθελοντικό σύστημα καταχώρησης και δηλώσεως των συμφερόντων. Λοιπόν, ο δεντολογικός κώδικας κώδικα συμπεριφορά, ποια κράτη-μέλη έχουν συντάξει τέτοιου κανόνε συμπεριφορά όσον αφορά τι απαιτήσει περί ακαιρεότητα που καλύπτονται από κώδικε για να προσανατολίζουν τα μέλη. Ε, γενικά βλέπουμε ότι έχουμε σχετικά περιορισμένη εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων και ο Γιάννους και ο Ντέιβιτ νομίζω ότι αναφέρθηκαν στο τι λειτουργεί, πώς πάει η εφαρμογή των μέτρων Έχουμε κάποια κράτη-μέλη ε, που έχουν ε, σημαντική ιστορία κώδικα συμπεριφοράς όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, η Πολωνία, εμπειρία 10, ίσως και 20 ετών. Στα περισσότερα κράτη-μέλη έχουμε σχετικά περιορισμένη εμπειρία όσον αφορά την χρήση αυτών των κανόνων και των κώδικων. Ε, τι συμπεράναμε εξετάσαμε τις αξιολογήσεις των συστημάτων και ρώτησε διάφορα κράτη-μέλη που συμπεριλαμβανόταν στην έκθεση Γκρέκο και ήταν τροφή προσκέψη τι πτυχές θα ενέπνεαν ενδεχόμενες μελλοντικές αναθεωρήσεις και αλλαγές ε, του κώδικα συμπεριφοράς των κρατών μελών. Ομάδες εργασίας κρατών μελών εξέτασαν διάφορα ζητήματα, τα συζήτησαν. Θέλαμε να δούμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, τι απαιτείται για να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη το κοινό στο σύστημα. Πρώτη ερώτηση, γιατί θέλουμε μεγαλύτερη ακαιρεότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια. Έχουμε ωφέλη, διότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη του κοινού, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και διοικητικός μηχανισμός για να ελέγχει τις δηλώσεις φερόντων, για να αποταμιεύει τις, τις ε, πληροφορίες και να δίνει προσανατολισμό τους στους βουλευτές. Τι θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί, πώς θα το προσεγγίσουμε. Ε, πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα. Θέλαμε να δούμε ποια είναι η εμπειρία που είχε αποκομιστεί, τι λειτουργεί. Να μεταθέσουμε την εμπειρία σε διαφορετικά πλαίσια. Να δούμε πού χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. τι ερωτήσεις θέτουν οι ευρωβουλευτές στη Συμβουλευτική Επιτροπή σας. Πού χρειάζεται περισσότερος προσανατολισμός, περισσότερες συμβουλές. Πώς θα το προσεγγίσουμε. Χρειάζεται ενεργή ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη. Κυρίως με τα κράτη-μέλη που πρόσφατα έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις των συστημάτων αυτών. Μετά τις λεπτομερείς συστάσεις του Γκρέκο. Έχουμε Ολλανδία, Σουηδία, διαφορετικά παραδείγματα που δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας για να εξετάσουν τις συστάσεις και να δουν πώς πρέπει να κάνουν τις δέουσες μεταρρυθμίσεις. Καμιά φορά υπήρξε επαφή και με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις συστάσεις. Έχουμε και διαφορετικές εθνικές παραδόσεις βλέπετε. Και θέλουμε μια προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο στις αξίες και υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα που στηρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους. Κάτι σημαντικό. Οι κώδικες συμπεριφοράς και συστήματα ακεραιότητας, όχι μόνο για κυβερνήσεις, αλλά και τον εκτελεστικό κλάδο, θεσπίζονται όταν ήδη τίθεται θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σκάνδαλο ξεσπάει. Και υπάρχει αντίδραση σε αυτό. Αυτό όμως δεν κλονίζει την εμπιστοσύνη του κοινού. Καλύτερα λοιπόν κανείς να προλαμβάνει. Συνεχώς να ελέγχει την κατάσταση. Και αυτό βλέπουμε στα κράτη-μέλη ότι υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια, μια μόνιμη ομάδα εργασίας που αξιολογεί τα θέματα αυτά, εξετάζει την υλοποίησή τους και πώς λειτουργούν οι διάφοροι κανόνες και τι αποτελέσματα έχουν. Εντάχει, δεν θα έλεγα ότι είναι συστάσεις. Θα έλεγα ότι είναι τομεί που θεωρούμε ότι μία αναθεώρηση των ισιόντων στα κάτι μέλη ίσως να εμπνεύσει προβληματισμό στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή, τι μπορούμε να εξετάσουμε εδώ. Όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς του Ευρωκοινοβουλίου, τι μπορεί να βελτιωθεί. Λοιπόν, στις δηλώσεις συμφερόντων. τακτικά δηλώνονται τα στοιχεία ενεργητικού και όχι τα χρέη. Οι περισσότεροι κανόνες θέλουν να εντοπίζονται και τα χρέη. Υποχρεώσεις. Όσον αφορά το εισόδημα των μελών του Κοινοβουλίου. Πόσο λεπτομερής πρέπει να είναι η δήλωση. Συζητείτε στη Γερμανία. Υπάρχει ένα παράδειγμα. Εδώ και δύο χρόνια. Μετά σύσταση Γκρέκο έγινε ιδέως αναθεώρηση και περισσότερα στοιχεία του εισοδήματο απαιτούνται και τα όρια έχουν αλλάξει το εισοδήματο. Δηλαδή από 250.000 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Μάλλον, συγγνώμη, από 2.500 ευρώ το μήνα και πάνω. Πολύ λίγες χώρες ε, το προσεγγίζουμε αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν όμως ε, κάποιες ε, προσεγγίσεις που είναι χρήσιμες να ληφθούν υπόψη όσον αφορά μετά της, για την κάλυψη των μελών της οικογένειας. Συζητείται στην Τρέκο το θέμα, πολλά κράτη-μέλη καλύπτουν και τα συμφέροντα των μελών της οικογένειας στις δηλώσεις, άλλες χώρες όχι. Η Γκρέκο συνέστησε ότι αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά να μην δημοσιεύεται, να μην δημοσιοποιείται. 12 κράτη-μέλη, αυτά που φαίνονται με σκοτεινό γαλάζιο, ε, απαιτούν να δηλώνονται και τα χρέη. Και με σκούρο χρώμα εδώ είναι τα κράτη-μέλη που ζητούν να καταχωρούνται και τα συμφέροντα των μελών της οικογένειας. Ε, τώρα, κατευθύνσεις, η δεύτερη συνιστόσα. Ίσως θα ήταν καλό να δούμε τι έγινε στη Σουηδία. Εκεί δίνεται ρόλος στη συνεχή μεταρρύθμιση και αναθεώρηση του συστήματος προστασίας ακαιρεότητος όσον αφορά τα επιφανή μέλη του Κοινοβουλίου. Και έπρεπε να δούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως με δύο παραδείγματα από χώρες εκτός αυτής όπου εκεί θεωρούμε ότι ίσως υπάρχουν παραδείγματα που μπορούν να μας εμπνεύσουν για στρατηγική για τα θέματα κυριότητος. Αυτό το είδαμε στην έρευνα συχνά. Δεν υπάρχει συνεχτική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό και ίσως χρήζει προβληματισμού. Για τον έλεγχο, την επιτήρηση, βασικό θέμα. Πώς το διοργανώνεις. Τα κράτη-μέλη ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον έλεγχο των δηλώσεων συμφερόντων. Στο τετράγωνο βλέπετε το Κοινοβούλιο, εσωτερικό έλεγχο και αυτοέλεγχο των μελών του Κοινοβουλίου. Έχουμε το σύστημα αυτό σε κάποια κράτη-μέλη, όπως στην Ολλανδία και στη Δανία. Κάμια φορά η δίκηση πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει και να ξεκριβώνει αν είναι σωστές οι δηλώσεις. Ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους τα κράτη-μέλη και ίσως εδώ το κοινοβούλιο ίσως να θέλει να το εξετάσει. Αν θα εξωτερικευτεί ο έλεγχος, θα ανατίθεται σε κάποιους φορείς ειδικού που αποκλειστικά θα ασχολούνται με τον έλεγχο των δηλώσεων συμφερόντων των μέλων του κοινοβουλίου. Αυτό ή κάτι ευρύτερο, όπως τον Καναδά. Φορέας με πολλούς πόρους που εξετάζει δηλώσεις των συμφερόντων των μελών του Κοινοβουλίου αλλά και όλων των δημοσίων ε, εκείνων που κατέχουν δημόσιες θέσεις και το ίδιο ισχύει και στην Ισπανία. Δεν φαίνεται εδώ στο σχήμα, σε πολλές χώρες έχουμε ε, συνδυασμό των προσεγγίσεων. Κάτι που επεκρίθη ευρύτατα, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι δηλώσεις συμφερόντων στις ε, σελίδες ε, σε διαφορετικές γλώσσες σε μορφή PDF. Είδαμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Τι συστήνει η Γκρέκο. Ο χάρτης σας δίνει εντάχει την κατάσταση. Σε κάποιες χώρες έχουμε παρόμοια συστήματα. Οι σκοτεινές χώρες σε χρώμα, στο σκούρο γκρίζο, έχουν ξεχωριστά έγγραφα. Κάποιες χώρες δίνουν ένα τεράστιο έγγραφο με όλες τις δηλώσεις που συμπεριλαμβάνονται, ενοποιημένες σε ένα έντυπο και κάποιες χώρες έχουν βάση δεδομένων που μπορεί να ερευνηθεί για συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένους βουλευτές, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κλπ. Τελευταίο θέμα, έλεγχος, επιτήρηση, το προανέφερα. Είναι σημαντικό να δούμε και ποιο είναι το διοικητικό κόστος η εξέταση προσεκτική απαιτεί και κόστος. Υπάρχουν φορείς με πολλούς πόρους σε κάποιες χώρες που εξετάζουν το πώς λειτουργεί το σύστημα ακεραιότητας του Κοινοβουλίου. Κάναμε μια ταχεία σύγκριση βάσει στοιχείων που μας έδωσαν τα κοινοβούλια. Δηλαδή, ποιος είναι ο αριθμός του προσωπικού που εργάζεται επί επεξεργασίας των δηλώσεων και το κοινοβούλιο ξεχωρίζει. Έχει πολύ μικρό αριθμό ατόμων που στηρίζουν την όλη διαδικασία. Μετά οι κυρώσεις. Ήδη αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι σε αυτό. Η έρευνα δείχνει και θεωρεί ότι ένας κώδικας συμπεριφορά ανευκυρώσεων είναι μια χαρτινή τίγρης. Δεν πείθει τον κόσμο και το κοινό θα πρέπει να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα σύστημα επιβολής κυρώσεων για να εμπιστευτεί το σύστημα. Ένα παραδειγματάκι. Στο δικό σας κώδικα συμπεριφοράς έχετε διατάξεις. Αναφέρονται αυτές στο πώς θα εφαρμόζει ο πρόεδρος το σύστημα των δηλώσεων συμφερόντων. Πώς θα ζητά από τη συμβουλευτική σα επιτροπή να εξετάζει με συγκεκριμένη δήλωση, αν δεν υπάρχουν διατάξεις που θα εξετάζουν τι γίνεται με τον πρόεδρο τα μέλη τη Βουλευτική Επιτροπή. Υπάρχει διάταξη αυτή στη Γερμανία από αυτού. Και είναι το σημαντικότερο σημείο. Πώ θα γίνει η αξιολόγηση της παράβαση των απαιτήσεων και των κανόνων. Και η έρευνα και η Γκρέκο επιχειρηματολογούν κατά του ελέγχου από ομοτήμους διότι οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων και καλύτερα να γίνεται αξιολόγηση ανεξάρτητη των ενδεχομένων παραβάσεων. Τέλος, άλλος τομέας, όπου ίσως χρήζει προβληματισμού, υπάρχει ετήσια υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς των μελών του Κοινοβουλίου. Το ξέρω αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη και τρίτες χώρες που ε, αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για την αξιολόγηση των επιδόσεων τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια τους χάρη στον Καναδά. Γίνεται εξωτερική αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων ακαιρεότητας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον κύριε Μπλομάγερ. Έχουμε τώρα χρόνο για συζήτηση και όταν περατωθεί η συζήτηση, αν ο Σβέν Κίγκολτ συμφωνεί, ε, θα του δώσω το λόγο. Εκτός αν Σβέν θέλεις τώρα το λόγο. Γκίγκολτ. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Δεν είναι ότι θέλω τόσο πολύ να συζητήσω, αλλά να κάνω κάποια ερωτήματα. Πρόεδρος, ωραία, ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις τότε. Θέλατε το λόγο. Ρίτσαρντ, Ρίτσαρντ Κόρμπ. Έχω ένα τεχνικό ερώτημα, αλλά μάλλον είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε με τον Σβέν. Πρόεδρος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ο Σφέν. Ναι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγητής θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις κυρίους για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Διαβάζοντας τις εκθέσεις και ακούγοντάς σας έχουμε μάθει πολλά. Θα ήθελα να πω πού βρισκόμαστε σύντομα. Όπως είναι προφανές, περιμέναμε τις μελέτες αυτές, διότι η σύνταξη μιας έκθεσης χωρίς να έχουμε τον προτέρων στη διάθεσή μας ε, τις εκθέσεις δεν θα ήταν και ό,τι πιο καλό, άρα έχουμε τώρα τα αποτελέσματα. Επίσης ε, έχουν δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα μου οι πρώτες συστάσεις για τις οποίες ε, μπορούν να διατυπωθούν δημοσία σχόλια. Και οι σκιώδεις βέβαια έχουν πρόσβαση. Αφού και οι σκιώδεις λοιπόν συμμετάσχουν, μετά θα υποβάλουμε την έκθεσή μας έχοντα λάβει υπόψη τα δικά σα πορίσματα και τι δικέ σα συστάσει. Θέλω να πω ότι είναι προσδεκτά ε, και τα σχόλια του κοινού. Αυτό μπορεί να γίνει απευθεία στην ιστοσελίδα και θα ήταν πολύ θετικό. Παροτρύνω τους πολίτες να συνεισφέρουν. Ερωτήσεις προς τον συνάδελφο από τον ΩΣΑ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συσχέτιση μεταξύ εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο έχετε δει και το θέμα της αντίστροφης σχέση του reverse causality, δηλαδή ισχύει ότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη όταν υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ή είναι πιο ε, διαφανή τα συστήματα, τα πολιτικά που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αξιοπιστία. Επίσης, τα αποτέλεσματα του κύριου Κοέν και τις συστάσεις του της άξαν πολύ μεγάλη προσοχή. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον ε, σε διεθνές επίπεδο έχετε βρει παραδείγματα για κοινοβούλια ή κυβερνήσεις διοικήσεις που στο σύστημα περί ομάδων συμφερόντων και ομάδων πιέσεων έχουν ε, θεσπίσει κανόνες όπως εσείς ε, ε, προτείνετε για την εκπροσώπηση των διαφόρων συμφερόντων. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι είναι κρίμα το γεγονός ότι το νομοθετικό ίχνος, το νομοθετικό αποτύπωμα χρησιμοποιείται τόσο σπάνια. Στο 2 όμως λέτε ότι θα μπορούσε ε, να υπάρχει ένας περιορισμός στον αριθμό διαπιστευμένων ατόμων αναοργάνωση. Έχετε παραδείγματα όπου οι χώρες λαμβάνουν ενεργά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη εκπροσώπηση των διαφόρων συμφερόντων στην νομοθετική διαδικασία, διότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες. Εσείς λέτε πιο αδύναμες θέλετε να χρηματοδοτούνται γιατί η οργάνωση είναι πιο δύσκολη. Εσείς σας πάρει ένα. Το Κοινοβούλιο και οι φορείς της Ένωσης ε, ακολουθούν την πρακτική αυτή σε κάποιους τομείς. Εσείς έχετε βρει στις μελέτες σας τομείς όπου θα ήταν σημαντικό κάτι τέτοιο. Αυτός γενικές παρατηρήσεις. Εν τέλει, θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το που αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την συλλογή δεδομένων. Θα με ενδιαφέρει συγκεκριμένα να μάθω πόσο βρήκατε διαθέσιμα δεδομένα για τη δραστηριότητα των λόμπι στο Συμβούλιο και στην Κομισιό, αλλά και ε, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Θα ήθελα να πείτε τι όρια σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων διαπιστώσετε ότι υπάρχουν τι περιορισμοί και αν μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο και για τη διαφάνεια που επετεύχθη τι βαθμός διαφάνειας επετεύχθη κάποιες ομάδες συμφερόντων βλέπω ότι επηρεάζουν το νομοθετικό, τις νομοθετικές προτάσεις και μάλιστα από πολύ πρόωρο στάδιο. Κάποιες άλλες ομάδες όχι. Αυτό μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία ήταν αυτά που είχαν να κάνουν με τα δικηγορικά, τις δικηγορικές ενώσεις, δικηγορικά γραφεία κτλ. Η ΜΚΟ φαίνεται ότι ψώνει τη φωνή τους μόνο όταν πλέον τα πράγματα έχουν δημοσιοποιηθεί. Μήπως πρέπει να δώσουμε κίνητρα ώστε όλοι να ακούγονται σε πιο πρώιμα στάδια. Τέλος. Δεν κατάλαβα και πολύ καλά, κύριε Μπλόμαϊερ, για αυτή τη βάση δεδομένων που αναφέρατε. Τα δεδομένα γκρέκο ουσιαστικά δηλαδή, έτσι. Όταν δεν υπήρχαν πρόσφατα δεδομένα γκρέκο, τι γινόταν δεν τα λαμβάνετε ε, στην έκθεσή σας. Υπόψη, ναι ή όχι. Επίσης, η επιλήρης δέσμη των κρατών μελών. Θα ήταν ενδιαφέρον αν είχατε ε, εξετάσει το σύνολο των κρατών μελών. Γιατί βλέπω για παράδειγμα ότι η Κροατία που όπως βλέπετε και σε κάποιο κομμάτι των δεδομένων και από ό,τι μαθαίνουν είναι από τα κράτη που πραγματικά έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος ε, όσων θα θέλαμε να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. δεν τα βρίσκω εδώ αυτά τα στοιχεία, αλλά θα ήθελα να μου πείτε γιατί δεν ήταν καθόλου εφικτό να έχετε την πλήρη δέσμη δεδομένων για τη σύγκριση. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο αυτό. Αυτά ευχαριστώ. Very Uh... Σας ευχαριστώ. Ρίτσαρτ, έχεις και εσύ ερώτηση και ο μετά. Ναι, το περίμενα ότι ο Σβέν. Και όντως με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό, άρα θα περιοριστώ μόνο σε κάποια τεχνικά ζητήματα. Στο 3 και στο 16 της εκθέσεως σας, που είναι νομίζω το ίδιο. Στο 3, σελίδα 14 και στο 16 της σελίδα 42 στην έκθεση Πώς κάνατε την κατανομή ανά επιτροπή, σε τι στηριχθήκατε. Στις ίδιες τις δηλώσεις ε, αυτών που πάτε στο ερωτηματολογιό σας, στο Μητρό του Κοινοβουλίου, απαιτείται εκεί να σημειώσει κανείς ε, σε ποια επιτροπή ενδιαφέρεται να έχει παρουσία. Άντρε. Ευχαριστώ πολύ Τζούτζι και όλους τους ε, παρόντες για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και αναλύσεις ε, της εκθέσεως που θα μας βοηθήσει στην εκθέση του συναδελφού Γκίγκολτ και όλων μας βέβαια που είμαστε Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε περισσότερο είναι το, ο βαθμός ανταπόκρισης στις ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές για την πρώτη μελέτη, την πρώτη έρευνα. Έγινε επανλήθευση με το Μητρό Διαφάνειας. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για μένα, για να αντιληφθώ την ε, χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του μέτρου, του Μητρώου Διαφάνειας. Επίσης, όταν λέτε ότι εμείς ως Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία των ομάδων στις επιτροπές που έχουν χαμηλότερη εκπροσώπηση αυτές. Ε, πώς το εννοείτε. Γιατί είμαστε πατέβαστοι ε, εάν πρέπει να προτιμούμε την συμμετοχική ή την ε, ε, κατεκπροσώπηση στην δημοκρατία, αλλά πάντως θα είναι χρήσιμο να δούμε αυτό που έχετε εσείς να προτείνετε. Για δε τις δηλώσεις των οικονομικών συμφερόντων, πολύ σωστά λέω Σβέν και το βλέπω και στην δική σας την έκθεση, καθώς ε, προέρχομαι από την τελευταία χώρα που μπήκε στην Ένωση, περάσαμε από πολύ αυστηρή ε, πολύ αυστηρό έλεγχο των ε, ζητημάτων της διαφθοράς, των σύγκρουσης συμφερόντων κτλ. Και κυρίως για όσους αναλαμβάνουν δημόσια καθήκοντα και δει ε, ως βουλευτές. Η Κροατία νομίζω είναι αυτή η οποία χρειάστηκε λιγότερες συστάσεις από την Επιτροπή Γκρέκο. Ευχαριστώ πολύ, Μαϊτέ. Ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα έχω να υποβάλω. Μελετήσατε μήπως το ζήτημα της έλλειψης ειλικρίνειας ε, στα βιογραφικά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τους τίτλους σπουδών, ε, ε, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση αυτών των πολιτικών ή των εκπροσώπων. τα στοιχεία που θα έπρεπε να ε, επαληθεύονται, ιδίω όταν μιλάμε για διαφάνεια. Γιατί θέλω να σα πω ότι στην Ισπανία δεν έχει γίνει μόνο μια φορά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι έχουν τίτλους και τελικά δεν τους έχουν. Δεν έχουν τα πτυχία αυτά που λένε. Για παράδειγμα, λέει κάποιος ότι έχει πτυχίο φυσικής από το Complutense και δεν ισχύει αυτό τελικά. Επίσης, ε, υπάρχει ε, το σύστημα προστασίας δεδομένων στην Ισπανία δεν μπορεί κανείς να πάει στο πανεπιστήμιο για να επαληθεύσει ότι πράγματι δεν έχει τον τίτλο, ότι δεν έχει το πτυχίο ε, το λόγο άτομο και έτσι εξαπατάται η κοινωνία και δεν μπορεί κανείς να επαληθεύσει τα βιογραφικά όλων αυτών των ατόμων. Το έχετε σκεφτεί, σας έχει απασχολήσει το ζήτημα. Μήπως θεωρείτε σωστό ότι θα έπρεπε να υπάρχει τελικά ένας οργανισμός που να έχει την αρμοδιότητα να επαληθεύει την ε, ύπαρξη ε, τίτλων, την κατοχή τίτλων, ε, εφόσον από τα πανεπιστήμια δεν γίνεται αυτό. Οι πολίτες όμως έχουν δικαίωμα να έχουν ακέραιους πολιτικούς. Δεν ξέρω, σας απασχόλησε αυτό και τι σκεφτήκατε σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, Αντινόλφη. Ευχαριστώ. Το συγγνώμη που απουσιάζει και ο Σκαστάλτο. Θέλω να ευχαριστήσω όμως τους εισηγητές. Έξοχη ήταν η παρουσίασή τους. Ενδιαφέρομαι πολύ όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κώδικα συμπεριφορά και το θέμα, το θέμα του λόμπι. Προέρχομαι από κίνημα πολιτών που και στο Εθνικό Κοινοβούλιο στην Ιταλία έθεσε το πρόβλημα των λόμπι που βρίσκονται ε, στα κέντρα εξουσίας και το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ σαν θέμα. Όταν μου έτυχε να εργαστώ στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Πολιτισμού που ανήκω εκεί, ξέρω τα θέματα όπως το copyright, μπορούσα για πρώτη φορά, είμαστε μια πολύ νέα αντιπροσωπεία, για πρώτη φορά ήρθαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είδα ακριβώς τι σημαίνει επαφή με τα μέλη των λόμπι. Και θα ήθελα και σε σελίδα μου στο διαδίκτυο ε, με ποιους ήρθα σε επαφή μέλη του, των λόμπι. Δεν σημαίνει ε, διότι η συνάντηση γίνεται με, και κλεισμένο των θυρών. Είναι όμως μια αυθόρμητη κίνηση, μια πρωτοβουλία δική μου αυθόρμητη, αυτή που έκανα, ούτω ώστε να να μπορούν να συμμετέχουν και εκείνοι που δεν μπορούν να μπουν στο κοινοβούλιο, αλλά να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι συμβαίνει στο κοινοβούλιο. Ασχολούμαι και με την ομάδα εργασία που εξετάζει τη μεταρρύθμιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου, μαζί με τον κύριο Κόρμπετ. Και είναι τιμή μου που ανήκω σε αυτή την ομάδα εργασία. Υπάρχουν πολύ επιφανή μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πεφωτισμένα μέλη. Στην ομάδα λοιπόν εργασίας τίθεται το πρόβλημα του κώδικα συμπεριφοράς και δυστυχώς παρά τις καλές προθέσεις φαίνεται ότι δυστυχώς η επιλογή της ομάδας εργασίας ήταν από ό,τι είδα και από ένα email ότι δεν εξετάζει τον κώδικα συμπεριφοράς. Δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις εκεί όσον αφορά τα δώρα που να δεχτούν οι βουλευτές ή όχι αλλά είναι πολύ θολά τα πράγματα όσον αφορά ε, τις διάφορε, την παροχή συμβουλών. Σε διαφορά με την προηγούμενη θητεία, το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη θητεία είναι να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το πρόβλημα. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα κανόνα που απαγορεύει σε κάποιον που έχει συγκρούσει συμφερόντων συγκεκριμένε να συμμετέχει σε εργασίες σαν μέλος μιας επιτροπής. Και θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήταν ένα μήνυμα για να πλησιάσουν οι πολίτες τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που πάντα τα βλέπουν με επικριτικό όμα. σε διαφορά, σε διάκριση με αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα εργασίας. Πρέπει εμείς εδώ να το αντιμετωπίσουμε το θέμα για να κάνουμε καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Α κάνω και εγώ λοιπόν μια ερώτηση. Και σας ξαναπάω πίσω κύριε Μπερτόκ στην αρχή της τοποθέτησης, της παρουσίασής σας. Με μια πιο θεωρητική μάλλον ερώτηση διορθώστε με αν ε, απατώμε, αλλά βλέπω ε, από την παρουσία σας ότι συνδυάζεται σαν σταθερές αξίες τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, ενώ είναι δυναμικές και αλλάζουν με, μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Άρα αυτό που θεωρείται ότι υπάρχει υποκειμενικά ε, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και χώρο δεν είναι δεδομένο και σε άλλη χρονική στιγμή και χώρο. Άρα θα πρέπει να προσαρμόζεται τα στοιχεία σας. Και ίσως θεωρήσετε ότι δεν ήταν το αναμενόμενο, αλλά εγώ από τις μελέτες που έχω δει και δεν είναι αρνητική απαραίτητα οι συσχετισμοί, αλλά όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο, όσο υψηλότερο το επίπεδο της διαφάνειας φαίνεται να και χαμηλότερο το επίπεδο της εμπιστοσύνης. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από την πολιτική κουλτούρα από την οποία προέρχεται ο καθένας. Δηλαδή, αν είναι υψηλό το επίπεδο της ε, ε καχυποψίας, ε, τότε μάλλον ε, όσο περισσότερη είναι η διαφάνεια, οδηγείται κανείς στη σκέψη ότι α, για να τα λένε τόσο πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά, θα πει ότι είναι πολύ βρώμικα όλα πίσω. Άρα λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω. Ε, τη γνώμη σας για το κατά πόσον ένας υπερβολικά μεγάλος ε, βαθμός και αριθμός πληροφοριών μπορεί να υπονομεύσει την ε, αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη. Πώς μπορούμε να βρούμε αυτή την ιεράρχηση των αξιών. Και εν τέλει, το πιο σημαντικό για μένα, είναι ότι διαφάνεια και lobbying έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης βιώνει το ζήτημα της εξουσίας. Δηλαδή είναι πολλές περιπτώσεις ε, που εγώ πιστεύω το όντι ότι η διαφάνεια όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά τους είναι και αντιπαραγωγική. let me open the floor to you. Uh... Ναι, θα σας δώσω το λόγο βέβαια. Να το πάρουμε ανάποδα, ο κύριος Μπλομάιερ πρώτος. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Για τον κύριο Κίκολτ και να διευκρινίσω τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε για τη μελέτη ήταν από δύο κατηγορίες με την υφιστάμενη έκθεση Γκρέκο όταν την πήραμε εμείς στα χέρια μας βέβαια κάπου στα μέσα Μαΐου, αρχές Ιουνίου άρα είχαμε στα χέρια μας όσες εκθέσεις Γκρέκο είχαν μέχρι τότε δημοσιευθεί επιπλέον αυτό κάναμε μια μελέτη με ερωτηματολόγιο που αποστήλαμε σε ευρωβουλευτές, σε όλους τους ευρωβουλευτές και σε διοικητικά όργανα τρίτων κρατών και άρα έχουμε συνδυάσει τα στοιχεία αυτά από τις εκθέσεις Κρέκο και τα ερωτηματολόγια χωρίς να είναι πλήρη σε όλα τους τα επίπεδα και τα στάδια για όλες τις χώρες κάποιες εκθέσεις ε, είχαν δημοσιευθεί από την Γκρέκο, άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτες και πληροφορίες από εκεί και χάρτες. Και κάτι άλλο, εκεί όπου δεν έχουμε πληροφορίες για κάθε κρατη κράτη-μέλη, μπορούμε νομίζω να κάνουμε τη διάγνωση με βάση την πορεία στην αναθεώρηση νομικού πλαισίου αλλά από την άλλη, από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτά που ορίζει το νομικό πλαίσιο και την πρακτική υλοποίησή του. Γι' αυτό και προτιμήσαμε να στηριχθούμε στις εκθέσεις Κρέκο, την επισκόπησή τους και βέβαια την συνομιλία με αυτούς που τους έχουν συντάξει. Κύριος Γκίκολτ. Πρόεδρε, μου επιτρέπεστε να επιμένω. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνω το εξής από τους πίνακες στην έκθεσή σα. Αντιλαμβάνομαι ότι μόνο χώρες για τις οποίες υπάρχει πρόσφατη έκθεση Γκρέκο καταγράφονται. Δεν βλέπω αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που απευθύνατε στα κράτη-μέλη. Πού θα τα βρω εγώ αυτά, τα αποτελέσματα, για το καθεστώς που επικρατεί ανάλογα με, τις, με τα ερωτηματολόγια σας. Ναι, λέει ο κύριος Μπλόμαϊερ, εκεί που βλέπετε κενό στον πίνακα, σημαίνει ότι το κράτος μέλος, το κράτος μέλος δεν απέστειλε απάντηση, δεν έχουμε πληροφορία για το σύστημα που έχει. Μη συγχωρείτε, <laughs> μπορεί, μπορεί να είμαι πράγματι πολύ χαζός, αλλά στο πίνακα υπαριθμών 5, σελίδα 25. Δεν βλέπω όλα τα κράτη-μέλη. Όχι μόνο κενά δηλαδή υπάρχουν, αλλά δεν έχετε καταγράψει ούτε καν τα κράτη-μέλη στο σύνολό του. Και αυτό το βλέπω σε όλου του πίνακε. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχετε 28 γραμμέ στο πίνακα. Μπλομαίρο. Ο αριθμό των κρατών μελών που βλέπετε στον πίνακα σχετίζεται με το τι κάναμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ή κοιτάγαμε εκθέση Γκρέκο, κοιτάγαμε απαντήσει στα για, τα 20, για 20 περίπου στην κάθε περίπτωση. Οπότε εκεί που έχουμε απαντήσει με την έκθεση Γκρέκο για ένα συγκεκριμένο θέμα, τότε το σημειώνουμε. Ήταν σαφέστερο τώρα δεν, βάλαμε, δεν περιλάβαμε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί δεν είχαμε πληροφορίες και για τα 28 και δεν μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε εάν υπήρχε απέτηση από την νομοθεσία, αφού δεν είχαμε στοιχεία. Καλά, να μην σας κουράζω, αλλά παρακαλώ, θα ήθελα να συμπληρωθούν όλοι οι πίνακες, να είναι διαφανής η κατάσταση. Πού δεν απαντήσανε, πού εσείς δεν είχατε πληροφορίες, πού δεν ισχύει καθόλου κάποιο σύστημα. Γιατί για μένα έχει σημασία το να ξέρω εάν έμεινε κενή μία γραμμή ή ένα πεδίο γιατί δεν υφίσταται καθεστώς ρύθμισης ή γιατί δεν σας έστειλαν απαντήσεις. Και στη συνέχεια για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζω τι συστήματα έχουν τα κράτη-μέλη και τα 28 όμως. Δεν είναι για μένα καθαρός ο πίνακας. Γιατί δεν είναι όλα τα πεδία συμπληρωμένα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν είναι συμπληρωμένα και καθώς θα ήθελα να έχω πλήρης δυνατότητα να συγκρίνω όλες τις πτυχές του συστήματος για όλα τα κράτη-μέλη, θα ήθελα να είναι πλήρης οι πινάκες. Εδώ δεν είναι πλήρης. Ας μην ξεκινήσουμε τώρα ένα πινκ-πονγκ από τον ένα στον άλλον, ναι, αλλά βλέπω ότι δεν καλύπτονται όλες οι πτυχές όπως θα ήθελα. Richard returns just time. I'll answer Richard's first because it's a quick and... Να απαντήσω στον Ρίτσαρτ ε, γιατί είναι σύντομο. Μας δώσατε εσείς, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα δεδομένα. Τα έχετε βάσει των διαπιστεύσεων ε, από Στη δημοσία όμως δεν ήταν διαθέσιμα. Το ε, γραφείο ερευνών σας μας έδωσε, η υπηρεσία ερευνών μας τα έδωσε αυτά τα στοιχεία. Τώρα για να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα του Σβέν. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε τα νούμερα, τους αριθμούς για την εκπροσώπηση. Ε, να διευκρινίσω κάτι. Δεν είπα ότι ε, θα πρέπει να ε, είναι λιγότερες οι ομάδες. Η δημοκρατία χρειάζεται πολλές ομάδες διαφορετικότητα και σίγουρα χρειάζονται πολλές ομάδες συμφερόντων για ανταλλαγή πληροφοριών, για να υπάρχει ανάλυση περισσότερων δεδομένων. Μετά όμως ε, ερωτώ, μπορεί να υπάρξει επαρκή δυνατότητα ανάλυση όλων αυτών των πληροφοριών και όχι υπερφόρτωση. Εγώ είπα ότι ορισμένοι ε, οργανισμοί έχουν πάρα πολλά άτομα διαπιστευμένα, άλλε λόγω πόρων έναν για παράδειγμα μόνο. Κάποιε οργανώσει επίση έχουν και πολλού τομεί πολιτική. γι' αυτό χρειάζονται και πολλά άτομα, Κάποιε άλλε όχι. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό να δούμε γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί διαπιστευμένοι που έρχονται στο Κοινοβούλιο και μετά να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε κατά πόσον ε, η οργάνωση Χ, παράδειγμα χάρη, θα πρέπει να έχει 10 διαπιστευμένους, ενώ ε, ουσιαστικά ασχολείται με ένα θέμα. Αυτό εννοούσα, αυτή ήταν η λογική μου. λέει ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε εκτάσει ενδεχόμενο να θεσπίσει όριο για τον αριθμό διαπιστευμένων ανοργάνωση ή ανα είδος οργάνωση. Αυτή είναι η ανα είδο οργανωσης αυτη ειναι η συσταση σας, υπάρχουν δύο. Άλλα λέτε όμως τώρα. Λέμε ε, professional consultancy, δηλαδή επαγγελματικά ε, γραφεία συμβουλευτικής σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο τώρα, δεν γνωρίζω κατά πόσο κάποια εθνική κυβέρνηση έχει επιβάλει, δεν ξέρω, μπορεί να με διορθώσει ο Γιάννους, έχει θεσπίσει όρια για τον αριθμό των ατόμων που να συμμετέχουν. Θα μπορούσα να πω όμως ότι ε, με εξαίρεση στη Βόσικτον εδώ υπάρχουν περισσότεροι ομάδες συμφερόντων και λομπίστες σε απόλυτα νούμερα. Ξέρω γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Άρα πρέπει και είναι νομίζω λογικό να ε, σκεφτείτε και τα περί προσβασιμότητας, ε, περί συλλογής τόσο πολλών πληροφοριών και το κατά πόσο μπορείτε μετά να τις επεξεργαστείτε αυτές τις πληροφορίες. Ε, και ναι, μπορείτε να έχετε πολλούς που έρχονται, αλλά να μπορείτε να τα αξιολογήσετε καλύτερα όλα αυτά. Για τη διευκόλυνση για τις ε, μη κυβερνικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών. Δεν θέλω να, ε, να υπαγορεύσω τι πρέπει να κάνετε στον ένα στον άλλο τομέα. Ουσιαστικά για την Κομισιόν πιο πολύ ε, αυτό που είπα. Ε, θεωρώ ότι δεν έχουν ε, οι, αυτές οι ομάδες ε, του ίδιου πόρους σε σχέση με τις ιδιωτικέ συμβουλευτικέ ομάδες. Θα έπρεπε ίσως να μπορέσει να δευκολύνεται τις ε, διαβουλεύσεις ίσως με χρηματοδότηση του ταξιδίου για να μην πηγαίνουν μια στην Κομισία, μια στο Κοινοβούλιο. Και είδατε και από τα δεδομένα ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς πολιτικής όπου δεν υπάρχουν πολλοί. Μπορεί να μην υπάρχει, όχι καθόλου, αλλά πάντων λιγότερο δημόσιο ενδιαφέρον ή ενδιαφέρον από πλευρά ε, ΜΚΟ. Ενώ ε, σε άλλε πολιτικές πρέπει να βλέπετε κάθε φορά, θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο ευρεία διαβούλευση. Το θέμα είναι να έχετε δυνάμει κάποιους πόρους ε, για να διευκολύνεται αυτές τις επαφές ε, και η πολιτική, η συγκεκριμένη, ο τομέας πολιτικής δηλαδή θα μπορούσε να αποφεληθεί αυτών των ευρύτερων διαβουλεύσεων. Πάντως έχει κάνει θετικά, έχει πάρει θετικά μέτρα η Κομισιόν για να διευρύνει ε, τις διαβουλεύσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άσκηση επιρροής τα στοιχεία για τις ΜΚΟ είναι ενδιαφέροντα. Αν δείτε τον πίνακα 4, στην ε, σελίδα 64, τις διαφάνειες που σας έχουμε δώσει, εγώ δεν έλεγα ότι δεν επηρεάζουν οι ΜΚΟ. Οι βουλευτές που συμμετείχαν στην έρευνα και αν μελετήσετε και δείτε τα ε, κόκκιν, τις κόκκινες κουκίδες, ε, λίγο ή αρκετά επηρεάζουν είναι το 16%. Δηλαδή θεωρούνται σημαντικός ε, συνομιλητής ή ΜΚΟ. Τα θέμα είναι η συχνότητα. Έρχονται σε τακτά διαστήματα και ε, είναι δραστήρια, συμμετέχουν δραστήρια σπορτικές. Είναι ε, ε, θεμητοί και σημαντικοί εταίροι. Αλλά όταν είναι εκεί, εκεί είναι το θέμα. Τι είναι ενδιαφέρον πάλι στον κύκλο της πολιτικής. Σελίδα 63 εκεί που παρακολουθούμε το κύκλο της πολιτικής. Υπάρχουν διακοιμάσεις το ποιος έρχεται, ποιος δεν έρχεται. Πάλι έχει να κάνει αυτό με τους πόρους. Κάποιοι ξεκινάνε στο σημείο α και φτάνουν μέχρι το ω, γιατί υπάρχουν οι πόροι για την παρακολούθηση μέχρι τέλους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν θα δουν σημαντικό όλα τα σημεία του κύκλου της πολιτικής, απλά υπάρχουν άλλα ζητήματα, άλλε παράμετροι και βέβαια υπάρχουν κάποιε οργανώσει που όπω τα Think Tank και ομάδε προβληματισμού μπορούν να πούν πιο πολλά πράγματα στην έναρξη, στην αρχή τη διαδικασία και όχι τόσο στην ε, φάση ε, της ε, τελικής επεξεργασίας ε, ενός νομοθετήματος. Υπάρχει δηλαδή μια διακύμανση στο τι μπορεί να συνεισφέρει ε, ο ΜΕΝ και ο ΔΕ. Διατύπωση, υλοποίηση το ένα άκρο και το άλλο δηλαδή του κύκλου πολιτικής. Και αυτό ισχύει παντού, σε οποιαδήποτε χώρα ε, υπάρχει αυτή η διακύμανση ε, της συμμετοχής και των αναγκών, ανάλογα με το ποιο σημείο, στο, στο, στο, στο ποιο σημείο του κύκλου πολιτικής ε, βρισκόμαστε κάθε φορά. Εσείς είπατε ποια ήταν τα ποσοστά απάντησης, νομίζω στην έρευνα και η γενική βεστιτοποίηση. Κοιτάξτε, 71 απαντήσεις είχαμε μόνο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό ότι δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση ή ήταν όλοι τόσο πολύ πολύ άσχολοι γιατί τους ασκούν ε, πιέσει αυτοί οι 2.000 λομπίστες, δεν ξέρω. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Και ο αριθμός ε, των ε, ακαδημαϊκών ερευνών, λέει ο κύριος Κόρμπετ. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση και γίνονται αντιληπτά τα υπέρ ε, όπως φαίνεται από τον τελικό πίνακα, ότι δηλαδή μπορεί ο κόσμος να κρίνει και να δει ότι πράγματι βελτιώνεται η διαδικασία λήψης των πολιτικών αποφάσεων και χάραξης πολιτικών. Και για να τελειώσω μια θετική νότα, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πράγματι μία από τις πιο ανοιχτές διαφανείς πολιτικές οργανώσεις ε, σε σχέση με όσες έχω μελετήσει και εξετάσει και διάφορους τομείς ε, πολιτικής. Νομίζω αυτά και μπορώ να δώσω τώρα το λόγο στο Γιάννος. Perdone, la, la pregunta sobre la falta de honestidad. Ναι, το ερώτημα όμως για την έλλειψη ειλικρίνειας ε, στα βιογραφικά των βουλευτών. Είπα, αν είχατε ε, ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γιατί σας είπα ότι σε κάποιες χώρες όπως είναι η Ισπανία δεν έχουμε νομικά τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε τους τίτλους που ισχυρίζεται ότι κατέχει ένα άτομο. I, I would... Καλώς. Ε, δεν το αναλύσαμε αυτό τα βιογραφικά των ε, Ευρωβουλευτών. Θεωρώ καλή την πίστη ότι τα βιογραφικά είναι πραγματικά και οι βάσεις και οι γνώσεις των ατόμων. Αν δείτε στις επιτροπές, Θέλαμε να δούμε ποια είναι η προγνωμοσύνη, αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, διότι ήταν πολύ νέο το κοινοβούλιο τότε για, την προηγούμενη θητεία. Μάλλον εδώ, αν είχαμε κάνει την έρευνα στι αρχέ θητεία του Κοινοβουλίου, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ποια είναι η εμπειρία, η τεχνογνωσία των ευρωβουλευτών που είναι εισηγητέ και όδη εισηγητέ κλπ. Αυτό θέλαμε. Ποιε είναι οι γνώσει του για τον τομέα που εξετάζουν. Διότι κάνει τη μεγάλη διαφορά αυτό. Πώς μπορεί να κατανοήσουν τις ε, εισερχόμενε πληροφορίε από τις ομάδες συμφερόντων υπάρχει αλλαγή, διακύμανση διότι συμμετέχουν διαφορετικοί βουλευτές σε κάθε θητεία, πολλοί βουλευτές είναι διαφορετικοί και κάποιοι παίρνουν διαφορετικά θέματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμική μνήμη ούτως είπε. μια συνέχεια σε κάθε επιτροπή για να γίνει ανάλυση πολιτικής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική σύσταση. Κανένα άλλο γνωστό πολιτικό σύστημα θα επέτρεπε τέτοια ανανέωση και νέα σκέψη και νέα προσέγγιση σε κάθε θητεία κοινοβουλίου. Όταν γίνεται η αλλαγή στη ΣΥΠΑ υπάρχει η δημόσια υπηρεσία και έχετε το ίδιο και στη Βρετανία, στα διάφορα υπουργεία μονίμους υπαλλήλους που μένουν όλη τη ζωή εκεί και γνωρίζουν τα θέματα. Τα όσον αφορά τα βιογραφικά, Απλώς εμπιστεύομαι αυτά που λένε τα βιογραφικά. Η πιο δύσκολη ερώτηση και θέμα. Πώς γίνεται συσχετισμός αιτίου και αιτιατού. Έχουμε ελάχιστα στοιχεία. Θα παραθέσω συγκεκριμένα παραδείγματα πρόσφατα και ιστορικά, παλαιά άμα δείτε πηγαίνει σε διαφόρους υπήρους. Στον πρόεδρο της Χιλής, τον πρόεδρο του Μεξικού, απέναντί τους υπάρχει μεγάλη μείωση εμπιστοσύνης λόγω της όλης ιστορίας στις χώρες αυτές. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο είναι ορατός πάντα. Και έχει διάρκεια, άμα υπάρχει ακυποψία από πλευρά του κοινού. Εδώ και ένα χρόνο, εδώ ο Καναδός υπουργό ε, αντιμετώπισε σκάνδαλο χορηγίας. Και μετά, εδώ και κάποια χρόνια μάλλον, και μετά δεν μπορούσε να ξανακερδίσει τις εκλογές στο κόμμα του. Τι λένε οι Ολλανδοί, υπάρχει ένα ρητό. Έρχεται με τα πόδια εμπιστοσύνη και φεύγει καβάλα, λέμε στην Ολλανδία. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνη, όταν αυτή απολεστεί, είναι κάτι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Εντοπίζουμε τους παράγοντες που δημιουργούν την εμπιστοσύνη και η διαφάνεια είναι ένας παράγον. Χρειάζεται και σφαιρική προσέγγιση και ένταξη η ποιότητα της πολιτικής, η παροχή υπηρεσιών, η ακαιρεότης παίζουν ρόλο. Εφαρμογή των κανόνων, σεβασμός των αξιών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπουμε την απαρχή της επιστημονικής έρευνας στον τομέα. Συνεργαζόμαστε όμως την προσπάθεια με στατιστικές υπηρεσίες των χωρών. Εντάχει τα άλλα θέματα, οι άλλες ερωτήσεις. Το θέμα της αποκαλύψεως στοιχείων. Όσο πιο υψηλή η θέση κάποιου, τόσο μεγαλύτερη διαφάνεια απαιτείται. Αυτή, αυτό δείχνει η εμπειρία. Αποκάλυψη οικονομικών συμφερόντων κλπ. Όμως, τι δείχνει η εμπειρία. Ότι δίνεται λιγότερη προσοχή στην εξακρίβωση να ελεγχθεί αν είναι πλήρες οι πληροφορίες. Το κάνουν τα δύο τρίτα των χωρών του ΩΣΑ, αλλά μόνο 16 με 17% των χωρών ελέγχουν, κάνουν εξακρίβωση του περιεχομένου των πληροφοριών. Γι' αυτό πολλές χωρές, όσον αφορά τους πολιτικούς κυρίως, ανοίγουν προς το κοινό, δημοσιεύουν τις πληροφορίες για να υπάρχει μια έλεγ, ένας έλεγχος από πλευράς του λαού του κοινού. Συμφωνώ με την Ιταλίδα συνάδελφο. Χρειάζεται ενεργή προσέγγιση. Να μην περιμένουμε. Είδαμε τι έγινε στην Ιταλία. Στις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τρία κύματα προσπάθειας θέσπισης νομοθεσιών για το λόμπινγκ. Δεν πρέπει να περιμένουμε. Μπορείτε να το κάνετε εσείς. Να παρέχετε πληροφορίες. Αυτή είναι η προσέγγιση και αυτό αναμένεται σήμερα που ζούμε στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ. Κατά τύχη, εγώ πρέπει να ευχαριστήσω τους τρεις εμπειρογνώμονες και τα μέλη για την άκρος ενημερωτική και χρησιμότατη συζήτηση. Πολύ τροφή προσκέψη. Θα τη χρησιμοποιήσουμε σε διάφορα πλαίσια, κυρίως στο πλαίσιο της εκθέσεως του κυρίου συγητού μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας και να είμαστε επαφή. Διότι θέλουμε να αντλήσουμε από το υλικό που διαθέτεται τους επόμενους μήνες. Επόμενη φάση θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Τίμερμαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλουμε όμως αυτή η επιθυμία να καθυστερεί τις διαδικασίες θα συζητηθεί το σχέδιο εκθέσεως την 19η Νοεμβρίου. Στόχος να ψηφίσουμε στην Επιτροπή αρχές του επομένου έτους και μετά να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Να πάμε στο επόμενο σημείο. Τελευταίο σημείο. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εντός του ΟΗΕ. Πώς να πετύχουμε καλύτερα τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε τον David McAllister που είναι συγγητής μας, που θα παρουσιάσει την όλη κατάσταση, που βρισκόμαστε επί του θέματος. Εξετάζουμε σχέδια συμβαστικών τροπολογιών σε αυτή τη φάση και σίγουρα μπορεί να μας διαφωτίσει από αυτού. Έχεις το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συναδελφοί, ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Η έκθεσή μου, τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ηνωμένα Έθνη. Είχαμε 10 από το ΕΛΚ, 7 από του Ελληνικέ Δημοκράτε, 9 από την ΚΟΕ, 5 από τους ΕΣΥΑΡ και 4 από την ΑΛΔΕ και του πράσινου και 2 από του EFTD. Συνολικά αυτέ ήταν οι τις οποίες το σύνολό τους ε, κρίνω όσο χρήσιμη και αξιόλογη συμπλήρωση στην έκθεσή μου. Εν γέννη συμφωνούμε πως ε, πρέπει να αποκτήσει μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο ΙΕΠΕΣ, ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Αυτό έχει να κάνει βέβαια κυρίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κονδύλια από πλευρά των κρατών μελών, γιατί σε τελευταία ανάλυση είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός του ΟΗΕ. Είναι λοιπόν απαραίτητο μεγαλύτερη διαφάνεια και ορατότητα των ποσών και της χρήσης τις οποίες την χάνουν αυτά στον ΟΗΕ. Το Κοινοβούλιο πρέπει τακτικά και σφαιρικά να κοιτάει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα και κονδύλια που διατίθενται για τη χρηματοδότηση του ΟΗΑ αλλά και συγκεκριμένων μέσων. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχα την επαφή με τους ε, σκιώδεις ηγητές, πλην ε, του εκπροσώπου της CCR, εκπροσωπήθηκαν όλες οι πολιτικές ομάδες. Ε, συνεργαστήκαμε για την επεξεργασία των συμβαστικών τροπολογιών, τις οποίες είχα έτοιμες μετά τις πρώτες προτάσεις. Από αυτές Έγιναν κάποιες συμπληρώσεις από την ΚΟΕ για κάποιες τροπολογίες σήμερα το πρωί. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε δηλαδή τις ε, συμβαστικές τροπολογίες ε, ώστε να ενισχύει τη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι σαφέστερη εικόνα των ευθυνών των Ηνωμένων του Οργανισμού των και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για τη συνεργασία, το ρόλο του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή της και ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας συμπληρωματικά προς τις ε, τροπολογίες αυτές, σοσιαλιστές, δημοκράτες και η ΓΚΟΕ ζητούν μια πρόσθετη συμβαστική η οποία θα αναφέρεται στην σύσταση μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί το πρώτο, το πρώτο βήμα για τον εκδημοκρατισμό των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η προσέγγιση προς ε, ένα κοινοβούλιο του κόσμου ε, νομίζω ότι είναι υπερβολική και δεν μπορώ να την ε, υποστηρίξω, άλλωστε νομίζω ότι και η ομάδα μου την ίδια έποψη έχει. Η κυρία Ταπαντέλ έχει ζητήσει την υποστήριξη γυναίκας υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ. Εδώ δεν εξασφαλίζεται ομοφωνία από πλευρά των εκπροσώπων των ομάδων. Αυτά για την έκθεσή μου. Ψηφοφορία τη Δευτέρα στην προσεχή συνεργασία μας και θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους σκιώδες συγκητές για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή μας. Όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, σύμφωνα με τον κανονισμό επιτρέπεται δύο ομάδες ή περισσότερες να αντικαταστήσουν τις ε, τροπολογίες τους με συμβαστικές και το κανονίσουν μεταξύ τους. Όσον αφορά την τροπολογία α που λέει στη σελίδα, κάτι προτείνεται από, από μία ομάδα. Εδώ έχουμε συμβιβασμό που προτείνεται τον εισηγητή, που ο εισηγητής εξετάζει όλες τις τροπολογίες και όχι μία τροπολογία του ΕΛΚ. Υποθέτω ότι τελικά εδώ έχουμε ένα λαφάκι στο έγγραφο, όπως παρουσιάζεται. Ο Γιώ Λάινεν πρώτα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μακάλιστερ για τις συμβαστικές τροπολογίες. Οι οποίες στόχο έχουν καταρχήν να προσδώσουν μεγαλύτερο ρόλο στα Οργανισμό Αθηνών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συντονίσουν καλύτερα τη συνεργασία των κρατών μελών έτσι ώστε να μιλάμε με μία φωνή στον κόσμο. Έχω υποστηρίξει και την ιδέα το κοινοβούλιο να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο, σαφέστερο ρόλο στον Οργανισμό Εθνών. Ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος ε, έχει όλο και περισσότερα θέματα να επεξεργαστεί, θέματα που ε, άπτονται της καθημερινής ζωής των πολιτών και πρέπει όχι μόνο η εκτελεστική εξουσία αλλά και η νομοθετική, τα νομοθετικά όργανα των κρατών από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν και όχι ως παρατηρητές όπως είναι η Διακοινοβουλευτική Ένωση. Γιατί παρατηρητές είναι και η Greenpeace και η Διεθνής Αμνηστία. Είναι παρατηρητές, ε, δεν έχουν κανένα καθεστώς αποφασιστικό, ενώ θα έπρεπε να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν βουλευτές των κοινοβουλίων είναι απλώς παρατηρητές. Ας ξεπεράσουμε την αλλεργία του ότι μια κοινοβουλευτική συνέλευση μετατρέπεται σε κοινοβούλιο του κόσμου. Δεν είναι αυτό. Απλώς λαμβάνουν τα εθνικά κοινοβούλια, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κοινοβουλευτικό ρόλο στην κοινοβουλευτική, σε μια κοινοβουλευτική συνέλευση των Εθνών. Συζητούν θέματα. Έτσι ξεκίνησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενημερώνονται, γνωμοδοτούν. Και εγώ θα ήθελα μια και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο φορές ήδη έχει απευθύνει έκκληση για μια κοινοβουλευτική συνέλευση στον, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μην δοθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι αναφέρεται σε ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο και οτιδήποτε άλλο ε, θα ήταν λάθος συμπέρασμα και κατακριτέο από τους επιστημονικούς και πανεπιστημιακούς κύκλους. Είναι μια κοινοβουλευτική συνέλευση αυτό που ζητούμε, περισσότερη διαφάνεια. Γιατί έτσι μπορούν και η αντιπολίτευση και όχι μόνο οι κυβερνήσεις να είναι παρούσες. Υπάρχει η δυναμική της πλειοψηφίας και όχι της ομοφωνίας με την οποία αποφασίζουν τα κοινοβούλια και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα βελτιώσει και τη σχέση με τον πολίτη από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Βλέπουμε ότι είναι πολύ μακριά από την καθημερινότητα των πολιτών. Και όταν βλέπει ο πολίτης ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς του ΟΗΕ, δεν θα ενδιαφερθεί ούτε εκείνος. Βλέπω ότι ενωμένη παραμένει αντίθετη στην πρόταση αυτή η αντιπροσωπεία του ΕΛΚ. Ελπίζω όμως να γίνει πιο δεκτική απέναντι σε κάτι το οποίο από κοινού έχουμε επαφασίσει στο παρελθόν. Ευχαριστώ κύριε Λάιεν, κυρία Ταπαράλλη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μακάλιστερ για την προσπάθεια που έκανε και τους άλλους όδους συζητητές που μίλησαν για τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Όπως τα γνωρίζετε πιθανότατα, εγώ είμαι εισηγήτρια για το S&D για την έκθεση αυτή, για την γνωμοδότηση. Ήδη συναντήθηκα με τον εισηγητή την περασμένη εβδομάδα και συμφωνήσαμε επί διαφόρων σημείων. Παρουσιάσαμε συμβαστικές τροπολογίες, δεχτήκαμε τις συμβαστικές ε, που προτάθηκαν τον εισηγητή στον αφορά τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΦΕΡΙΠΗΝ τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με τους διεθνείς φορείς. Επί δύο σημείων όμως δεν συμφωνήσαμε και εκφράζω τη θλίψη μου γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη δημιουργία με, με σε, ε, συνέλευσης ε, κοινοβουλευτικής στον ΟΗΕ. παρουσιάσαμε μια πρόταση, πρόταση τροπολογίας, μια συμβαστική τροπολογία και δυστυχώς δεν υπήρξε συμφωνία. Ελπίζω στο τέλος τελικά να επιτευχθεί μια συμφωνία από αυτού. Οι επιχειρηματολογίες ήδη παρουσιάστηκαν. Δεύτερο σημείο, όπου το είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αφορά την εκλογή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον κύριο Μπαρσό παρουσίασα μια τροπολογία που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει έναν Ευρωπαίο πολίτη, μια Ευρωπαία υποψήφια, μια γυναίκα για αυτή τη θέση. Απερίφθη από τον κύριο Μακάλιστερ αυτή η τροπολογία, όμω ζητώ παρόλα αυτά από τι άλλε πολιτικέ ομάδε την υποστήριξή του, ώστε να εκλεγεί μια γυναίκα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη θέση. Παρουσίασα μια προφορική τροπολογία που λέει το εξή και αγγλικά ζητά να υποστηριχθεί μια γυναίκα υποψήφια για τη θέση της Γενικής Γραμματέως και μετά θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε γυναίκες υποψηφίους ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους καταγωγή. Όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα για την υποστήριξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις ε, από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υποστηριχθεί η ισορροπία των φίλων Είναι μια πρόταση αυτή. Κατά βάθο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής των γυναικών. Θέλω όμως να πω ότι η ισότητα των φύλων είναι σημαντικότατη ε, αναφέρεται και στην έκθεση για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Νόμου είναι κάτι που αφορά τις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Πιστεύω ότι θα θέλαμε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, τις γυναίκες ούτως ώστε να αναλαμβάνουν ηγετικέ θέσεις. Ελπίζω και άλλες πολιτικές ομάδες να συμφωνούν με αυτή την πρόταση από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν άκουσα και βλέπω ότι υπάρχει συμφωνία. Αλλά θα σας ζητούσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να υποστηρίξετε την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει ψηφοφορία αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ ο κύριος Σόλτς. Um, ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω, αλλά ήμουν στην Επιτροπή Εμπορίου και συζητούσαμε κάποιες διαπραγματεύσεις και έπρεπε να επιλέξω πού θα παρίσταμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες από πλευράς ομάδας μας συμφωνούμε με τη διατύπωση θα θέλαμε να προσθέσουμε και κάποια ζητήματα που είχαμε θέσει στην αρχή και δεν έχουν συμπεριληφθεί αλλά ελπίζω ότι θα συμπεριληφθούν όλα και συζητώντας συμβαστικές θα πετύχουμε καλά αποτελέσματα τελικά. Διότι είναι πάντα περίπλοκο να αναφέρεται κανείς στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον ΟΗΕ. Να μην αναμειγνύει κανείς θεσμικά και πολιτικά ζητήματα. Να, να περιοριστούμε στην προσέγγιση που θέλουμε να προτείνουμε στην ΑΦΕΤ, στην καθήλια αρμόδια επιτροπή. Στηρίζω λοιπόν και εγώ και ομάδα μου η αδίποτε πρόταση επανεξετάζει τον θεσμικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον ΟΗΕ χωρίς ανάμειξη με τα πολιτικά προβλήματα που πρέπει να συζητηθούν στην Επιτροπή ΑΦΕΤ ή σε άλλες επιτροπές ε, όπως την Επιτροπή Ανάπτυξης. Δηλαδή, ε, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον ΟΗΕ. Ελπίζω στην επόμενη συνάντηση να προχωρήσουμε και στηρίζω αυτό που αναφέρθηκε. Για να μην εφαρμόσουμε και στο σύστημα το ΙΕ το θέμα της ισότητας των φύλων ε, ε, σε όλα τα κάτι μελη τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να στηρίξουν μια τέτοια υποψηφιότητα. θα πρέπει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημοκρατία όσον αφορά την ισότητα του φύλου. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται εκδημοκρατισμός όσον αφορά την, ε, ε, τη σωστή εκπροσώπηση της ε, κοινωνίας. Ζωζέ Μαρία. Τρία σημεία. μια γυναίκα να γίνει γενική δραματέας. Εξαιρετική η ιδέα σας πραγματικά. Όμως, αυτό θα ήταν μια πρόταση. Γιατί άλλοι φορείς μπορούν να κάνουν άλλες ή αντίστοιχες προτάσεις. Αν θέλουμε να ασκήσουμε δε κάποια αυτοκριτική, θα έπρεπε ίσως να ξεκινήσουμε να κάνουμε για το σώμα για το κοινοβούλιο μας αυτές τις προτάσεις. Δεν ξέρω αν θα πετύχει η πρόταση αυτή βέβαια. Μια εκλογή ναι μπορεί να πετύχει. Αυτό είναι το πρώτο. Δύο γυναίκες τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είχαμε ήδη, λέει ο κύριος Κόρμπετ. Ναι, είχαμε, λέει ο κύριος Τερικάμπρας. Εγώ λέω την πρόταση μια γυναίκα να είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι, αυτό δεν έγινε στις τελευταίες, ε, στις τελευταίες εκλογές και δεν νομίζω ότι θα γίνουν και στις επόμενες. Το αφήνουμε στους ψηφοφόρους ή όχι. Απράγματι είχαμε, έστω έχουμε καλύτερη εμπειρία δηλαδή από ό,τι στα Ενωμένα Έθνη εμείς. Πράγματι, έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε. Δεύτερον, η ανανέωση του σώματος, όπως τα είπε και ο Γιώλάινεν. Εγώ νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Κάτι πρέπει σίγουρα να γίνει και μάλιστα γρήγορα. Θα ήθελα ε, όμως να δημιουργηθεί ένα δεύτερο ε, που θα αντικαθιστά το μη αποτελεσματικό σώμα. Δηλαδή, αν ένα ε, σώμα, μια βουλή δεν είναι ε, αποδοτική, ε, αποτελεσματική, να έχουμε και άλλη μία που θα είναι δύο φορές αποτελ... επομένως πιο αναποτελεσματικό αυτό το σύστημα. Τώρα, στροπολογίαση πάρα πολύ σύντομα και ήπια αναφέρεται κάτι το οποίο εγώ πρότεινα και συγκεκριμένα ζητά μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι πολύ δέχομαι ότι αυτό που πρώτα μπορεί και να μην γίνει δεκτό. Ήθελα απλά να πω ότι δεν κάνω τέτοιες αόρισες προτάσεις. Ελαφρά την καρδία. Τι εννοώ όταν μιλάω για μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. σε σχέση με το βέτο. Νομίζω ότι θα ήταν πιο δημοκρατικός αυτός ο φορέας εάν το βέτο δεν εξαρτάται από έναν. Να είναι απαραίτητο, ναι, όπως είναι τώρα σε άλλους φορείς, σε άλλους οργανισμούς. Δύο-τρία βέτο. Θες πω, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Όλα να εξαρτώνται όμως από μία και μόνη χώρα είναι μεσαιωνικό κατά την άποψή μου αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. I give the floor. Ευχαριστώ. Ξανά ο εισηγητής για να απαντήσει. Έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα έδωσε καρπούς και έδειξε ότι συμφωνούμε επί πολλών σημείων. Επί τριών δεν συμφωνούμε. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το ρόλο της κοινοβουλευτικής συνελεύσεως του ΙΕ που εξαρτάται ανάλογα με τις διάφορες απόψεις υπάρχει συμφωνία, διαφωνία και τώρα γυναίκα υποψήφιος για γενική γραμματέας του ε, ΟΗΕ λάβαμε όλες τις τροπολογίες και από εσάς κύριε Σόλτς και από την ε, ΓΚΟΕ από αυτού και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Εγώ θα έλεγα δημοκρατικά τη Δευτέρα να ψηφίσουμε και τελικά θα καταλήξουμε μέσω ψηφοφορία σε κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πολύ λογικό ακούγεται αυτό. Και η ψηφοφορία πράγματι προβλέπεται την επόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Φοβόμαι ότι θα απουσιάζω. Έχουμε το συνέδριο του Εργατικού κόμματο που όπως τα ξέρετε υπάρχει αύξηση του αριθμού των μελών ανακάμπτει το κόμμα, θα χάσει τη ψηφοφορία. Σα εύχομαι όμω μια πάρα πολύ καλή συνεδρίαση, οπότε φτάσαμε στο τέλος της συνεδριάσεω. Η επόμενη τακτική συνεδρίαση είναι στις 28 του Σεπτεμβρίου, όπως προανέφερα, και επόμενη στις 22 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρα συνεδριάσεως. Γεια σας. Καλή σας μέρα.